Καλημέρα σας. Bonjour. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Παρακαλώ καθίστε. Θα συνεχίσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Θα περάσουμε αμέσως στις ψηφοφορίες και στη συνέχεια θα προβούμε σε μια ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο Φερέιρα πρώτη ψηφοφορία σήμερα το πρωί για το θέμα της απαλλαγής του 2018 Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Κούτα Γιάρ είναι η συγγήτρια, η Κούτα Ζάρ, μας παρουσίασε την εισήγησή της το Δεκέμβριο, 42 τροπολογίες υποβλήθηκαν και 10 συμβιβαστικέ τροπολογίες έγιναν αντικείμενο πολιτικής διαπραγμάτευσης μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Θα ήθελε η εισηγήτρια να προσθέσει κάτι πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, παρακαλώ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε, Πρόεδρε, τους συναδέλφους ε, για τη συμβολή τους, για τη συνεισφορά τους. Προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε στο κείμενο όσες περισσότερες συνεισφορές γινόταν ε, και να ικανοποιήσουμε τις διάφορες πολιτικές προτεραιότητες. Θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα όλους για τη συνεργασία τους. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Ε, περνούμε ευθύ αμέσω στη ψήφιση λοιπόν του κειμένου ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια θα περάσουμε στην τελική ψήφιση του κειμένου επί του συνόλου. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας. Ποιος είναι υπέρ. Θα ξεκινήσει η ψηφοφορία τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία με τις ηλεκτρονικές κάρτες. Ποιος είναι υπέρ. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ. Τέλος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η έκθεση. 31 ψήφοι υπέρ. Συγχαρητήρια. 35 ε, ψήφοι υπέρ, 31 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, 35 στο σύνολο, 0 αποχές. Σας ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ και συγχαίρω την εισηγήτρια. Περνούμε στο επόμενο κείμενο, ψηφοφορία για την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απόφαση του Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συντονιστές αποφάσισαν να συντάξουν γνωμοδότηση με τη μορφή επιστολής που ε, θα συντάξει ο πρόεδρος. Δεν υπήρξε αντίρρηση επί της διαδικασίας. Έχουμε μία μόνη ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ. Παρακαλώ. Πέρας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Περνάμε τώρα σε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα, γιατί περιμένουμε την Επίτροπο Ελίζα Φερέιρα για την ακρόασή της. Θέλω να σας πληροφορήσω και να σας πω ότι η ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε με την Επίτροπο ε, θα λάβει χώρα ως εξής. Καταρχάς θα δώσω το λόγο στο συντονιστή. Η Επιτροπή θα, ε, η Επίτροπος θα απο, απευθυνθεί ξεχωριστά σε κάθε έναν από τους συντονιστές και μετά θα δώσω το λόγο σε οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής μας θελήσει να τον πάρει. Θα καταγράψουμε τις ε, ερωτήσεις και η Επίτροπος θα απαντήσει ομαδικά ε, στις ερωτήσεις των, των μελών. Κάνουμε λοιπόν ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και... Ε, θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση όταν έλθει η Επίτροπος. Θα τα πούμε εντός ολίγου. Je Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Παρακαλώ καθίστε. Έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα κοντά μας στην Επιτροπή μας για τις Περιφέρειες και τα Περιφερειακά Θέματα την Επίτροπο κυρία Ελίζα Φερέιρα, αρμόδια για την Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στην Επιτροπή μας από την από την ε, αναέγκρισή σας ε, για το αξίωμα αυτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 27 ε, Νοεμβρίου. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας αυτό. Σας συγχαίρω επισήμως για την ανάληψη των καθηκόντων σας. Ε, θα περάσουμε πέντε χρόνια μαζί, θα δουλέψουμε μαζί εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι σημαντικές και Πρώτα απ' όλα το πιο σημαντικό είναι η οριστικοποίηση της διαπραγμάτευσης για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ειδικότερα για τον φάκελο και τα κονδύλια που ε, προβλέπονται για τους τομείς της αρμοδιότητάς μας. Έχουμε τον κανονισμό για τις κοινέ διατάξεις, για το ΦΕΝΤΕΡ, για το ΕΤΠΑ, όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά πρέπει και να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν, έτσι ώστε όλες οι περιφερειές της Ευρώπης σε εύλογο χρονικό διάστημα να έχουν τους αντίστοιχους κανονισμούς που τους χρειάζονται για τον προγραμματισμό τους για το εγγύς και απότερο μέλλον. Στη συνεδρίαση των συντονιστών αποφασίστηκε να παγώσουν μέχρι το, τις 27 Φεβρουαρίου οι, όλοι οι πολιτικοί τριμερείς διάλογοι. διάλογοι. Γιατί περιμένουμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ένα προπολογισμό που να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, που να αντιστοιχεί στο μέγεθος των προκλήσεων και που να μην θυσιάζει την πολιτική συνοχή. Περιμένουμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προσδιορίσει, να καθορίσει τη θέση του για το σύνολο ε, των άρθρων που ε, ε, εντάσσονται στον κανονισμό, ε, για τα οποία βέβαια έχουμε εμείς εντολή διαπραγμάτευσης και τα οποία δεν αποτελούν μέρος του κοιτίου διαπραγμάτευσης, του negotiating box και που ε, σύμφωνα με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνονται αντικείμενο συναπόφασης. Άρα έχουμε εξουσιοδότηση, έχουμε εξουσία ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε προνόμιο ως συνομοθέτες και αυτό πρέπει να γίνει απολύτως σεβαστό και να τηρηθεί ε, στο σύνολό του και 100%. Και λέγοντας αυτά ουσιαστικά εκφράζω κοινή θέση, ε, κοινή θέση εξ ονόματος όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι σαφής ο, ο προσανατολισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι καθορίστηκε στη διάσκεψη των Προέδρων των πολιτικών ομάδων στη σχετική συνεδρίαση εντό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό το λόγο, κυρία Επίτροπε, σήμερα ομόφωνα σα ζητούμε να δουλέψουμε μαζί βάσει του κανονισμού που προεβλέπει μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη του ΕΤΠΑ και του ε, ΦΕΟΓΑ ένα μεταβατικό κανονισμό για να υπερασπιστούμε τη συνοχή, να την προστατεύσουμε με ορίζοντα το 2021. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο στις διαπραγματεύσεις που επίκυνται, που έπονται σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα προϋπολογισμού, με θέματα δημοσιονομικά. Να ε, ε, στηρίξει αυτή τη θέση την οποία έχουμε επανειλημμένως υπερασπιστεί. Στις διαπραγματεύσεις, στις ανοιχτές, μπορούμε να καταλήξουμε στο βέλτιστο δυνατό κανονισμό, στο πιο ωραίο κείμενο αν όμως θυσιάζεται ο προϋπολογισμός, τελικά οι στόχοι της συνοχής θυσιάζονται. Και η Επιτροπή μας για, τα, για τις περιφέρειες και την περιφερειακή ανάπτυξη είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κονδύλια για τα οποία είναι αρμόδια. Ε, ο προπολογισμό που παρουσιάζει η Φιλανδική Προεδρία στο Συμβούλιο δεν είναι αποδεκτός για εμάς. Το έχουμε πει και το επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά σήμερα. Και εκφράζουμε και διατυπώνουμε ελπίδες για τις προτάσεις που ε, θα έρθει να καταθέσει στο τραπέζι η επόμενη Προεδρία. Σίγουρα αυτό το οποίο είναι αλήθεια σήμερα μπορεί να μην είναι αλήθεια αύριο και ελπίζω ότι θα κινηθούμε ε, ε, πέρα από αυτές τις γραμμές και ότι οι γραμμές αυτές θα οπισθοχωρήσουν. Η Επιτροπή μας είναι αρμόδια επί της ουσίας για να εξετάσει τον μηχανισμό για μια δίκαιη μετάβαση η οποία θα επιτρέψει τη συγκέντρωση κονδυλίων ε, σε ύψους 100 δις ευρώ ώστε να βοηθηθούν οι περιφέρειες ώστε να βοηθούν να βοηθηθούν οι περιφέρειες να, ε, να περάσουν αυτό το μεταβατικό στάδιο έτσι ώστε να φτάσουν σε μια οικονομική δραστηριότητα που θα έχει χαμηλές εκπομπές ε, ρήπων. Θεωρούμε, κυρία Επίτροπε, ότι σε αυτό το πλαίσιο η ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε με εσά σήμερα ε, είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Την περιμέναμε με μεγάλες προσδοκίες και με μεγάλη αγωνία. Τα μέλη της Επιτροπής μας έχουν πολλές ερωτήσεις να σας υποβάλουν συνολικά για το μέλλον της συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα για τον κανονισμό αυτό για την μετάβαση, τη δίκαιη μετάβαση προς μια οικονομική δραστηριότητα με χαμηλές εκπομπές ρήχων, ρήπων με μείωση κατά 5% ε, αυτών των εκπομπών. Θα ήθελα λοιπόν να ε, δώσω το λόγο στους συντονιστές. Θα σας ζητήσουμε να απαντήσετε άμεσα ε, σε κάθε συντονιστή και στη συνέχεια θα ανοίξει η συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής μας, με τους βουλευτές, οι οποίοι θα υποβάλουν διατυπώσεις και σχόλια, θα τα συγκεντρώσουμε ομαδικά και θα απαντήσετε στο τέλος ε, στις ερωτήσεις που θα έχουν θέσει τα μέλη της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής. Δίνω λοιπόν ευθύ αμέσω το λόγο στον κύριο Νοβάκοφ Εκτός και αν θέλατε εσείς, κυρία Επίτροπε, να πείτε δύο λόγια εισαγωγικά. Εάν όχι, περνάμε αμέσως στη συζήτηση. Δίνω το λόγο στον Αντρέη για το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητή Επίτροπε, θυμάμαι κατά την ακρόασή σας ως υποψήφια για τη θέση αυτή, για αυτό το χαρτοφυλάκιο, μέσα στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης, χρειαζόμαστε μία στεναρή επιτροπή. Τότε δεν γνώριζα ότι τόσο γρήγορα θα φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή. Σκέφτηκα ότι μέχρι την Κροατική Προεδρία ή στην απαρχή της Γερμανικής θα φτάσουμε σε ε, μία συμφωνία σε σχέση με τα ταμεία, ιδιαίτερα τα διαρθρωτικά και επενδυτικά. Δυστυχώς η αρχή του έτους μας απογοήτευσε. Δεν μιλώ εξ ονόματος ολόκληρης της Επιτροπής, αλλά θα ήθελα να πω ότι οι συνάδελφοι έχουν απογοητευθεί από την καθυστέρηση, η οποία δεν οφείλεται στο Κοινοβούλιο, αλλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στην Επιτροπή, αλλά στο Συμβούλιο όλοι μας είμαστε εκλεγμένα μέλη και βρισκόμαστε στις εκλογικές μας περιφέρειες σχεδόν κάθε εβδομάδα. Συνομιλούμε με τους ψηφοφόρους μας και οι πολίτες δεν κατανοούν γιατί έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ. Γιατί δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, γιατί το Συμβούλιο δεν έχει εντολή δεν έχει λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις. Υπάρχει ένα κουτί στο οποίο εισαγάγουμε στοιχεία, βγάζουμε μερικά και γι' αυτό το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δικαιολογώ τους πολίτες μας. Θα πρέπει να έχουμε ένα plan B, να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ε, πώς είναι δυνατόν να αναβάλουμε την ε, μεταβατική περίοδο του ε, ενός έτους σε σχέση με το πολιετές. Όποια και να είναι η απόφαση θα πρέπει να είμαστε θαρετοί και να εξηγήσουμε τη θέση μας, διότι υπάρχει ευροσκεπτικισμός, έκδηλος ευροσκεπτικισμός και Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις, δεν μπορεί να προχωρήσει. Έχουμε και άλλα θέματα προς αντιμετώπιση, γι' αυτό ας μην περιπλέκουμε και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, Αντρέη. Η Επίτροπος έχει το λόγο για να απαντήσει. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Νοβάκοβ, συνάδελφοι, πρώην συνάδελφοι, σας εύχομαι καλή χρονιά, καταρχήν. Δεύτερον, εκτιμώ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκομαι σε συνεχή επαφή με εσάς τους ευρωβουλευτές. Ως προς το θέμα που θίξατε, κύριε Νοβακόβ, νομίζω ότι όλοι συμμεριζόμαστε αυτή την ανησυχία με τα θέματα χρονισμού καθώς και τη διαδικασία για την ε, επόμενη περίοδο υποστήριξης. Έμαθα από την πρώτη παρέμβαση του Πρόεδρου της Επιτροπής ότι υπήρχε αυτή η διάθεση του Κοινοβουλίου, η πρόθεσή του να προχωρήσει. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος αυτό για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης, έτσι ώστε οι ευεργετούμενοι να μην στερηθούν από την πολιτική συνοχής, να μην υπάρχει ένας αποκλισμός. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό με κατέλαβε εξαπίνης αυτή η θέση, αλλά θα ήθελα να πω ότι με την ε, Γενική Διεύθυνση, με το προσωπικό και με εσάς θα προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος έτσι ώστε να μην πληγούν οι ευεργετούμενοι. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό, να δεσμευτώ με εσάς, έτσι ώστε να συνεργαστούμε όλες μας οι υπηρεσίες αλλά και εσείς και να δούμε πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε αυτό το αρνητικό κόστος προς τις περιφέρειες, τις ΜΜΕ, τις δημοτικές αρχές. Αλλά το θέμα είναι κατανοητό. Θα πρέπει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες επαρκώς. Αυτή είναι η απότερη ελπίδα μου. Ξέρετε πόσο μας απασχολεί αυτό το θέμα και τώρα οι συνομοθέτες, εμείς δηλαδή, θα πρέπει να συντονίσουμε τα τελευταία βήματα. Οι καταστάσεις έχουν ως έχουν. Δεν μπορώ να σχολιάσω ένα άλλο θεσμικό όργανο. Απλώς σας ευχαριστώ που συμμερίζεστε αυτές τις πληροφορίες. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο το στόχο της ίδιας μας της πολιτικής. Ευχαριστώ. Κωνσταντς ε, Κρέλ για τους σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Επίτροπε. Και σας ευχόμαστε μια καλή αρχή και σίγουρα δεν θα είναι εύκολο αυτό το έτος το 2020. Συμφωνώ με τις ανησυχίες τις οποίες εξέφρασε ο Ανδρέι Νόβακοφ όπως ε, τα είπε είναι τα πράγματα. Και μπορώ να πω με απόλυτη σαφήνεια ότι και την προηγούμενη φορά είχα την ε, χαρά αλλά και την ευθύνη τον τελευταίο κανονισμό να τον ε, δουλέψω το 2013 και 2014 και πραγματικά οι διαπραγματεύσεις ήταν σκληρές τότε δεν ήταν πιο απλές, αλλά τουλάχιστον ήταν δυνατόν να τύχουν διαπραγμάτευση σε στοιχεία τα οποία έχουν μπει πλέον στο κουτί των διαπραγματεύσεων και τα οποία καμία προεδρία δεν διατίθεται να συζητήσει. Αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα το δεύτερο ημίση του έτου, από το Σεπτέμβριο δηλαδή μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, θα έχουμε το χρόνο για να συζητήσουμε το 50% της πολιτικής συνοχής και να κάνουμε διαπραγματεύσεις. Μα δεν πρόκειται να προλάβουμε. Και αυτό επισημένοντας ε, το γεγονός ότι η πρόταση για το πολιτιστικό δημοσιονομικό πλαίσιο είναι μόνο κατά το ίμιση αποδεκτή. Δεν μπορεί λοιπόν να έχουμε μόνο την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειαζόμαστε πιο πολλά. Ε, μας κάνετε κι εσείς μια πρόταση για το Ταμείο α, Δίκαιης Μετάβασης και είπατε ότι θα χρειαστούν επιπλέον πόροι. Αυτό δεν έχει μπει σε καμία όμως πρόταση προς το παρόν. Και ως εκ τούτου πιστεύω ότι θα χρειαστεί μία μεταβατική περίοδος για την πολιτική συνοχή από το 2020-2021. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την Επιτροπή Γεωργίας έχει κάνει τα ανάλογα για την πολιτική γεωργία. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια κάποια βεβαιότητα ότι τα χρήματα αυτά, αυτά θα κρατεθούν το 2021 και πιστεύω ότι όλα αυτά θα πρέπει από κοινού να τα προετοιμάσουμε για την πολιτική συνοχή. Γιατί ακόμα και αν το πετύχουμε μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, 15 Δεκεμβρίου να ολοκληρώσουμε τι διαπραγματεύσει, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα είμαστε έτοιμοι από τον Ιανουάριο του 2021 να ξεκινήσουμε με την πολιτική συνοχή. Το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς οι ίδια ότι στην τρέχουσα περίοδο υπήρξε καθυστέρηση 1,5-2 ετών παρά το γεγονός ότι είχαμε ολοκληρώσει τα χρεώδη μέχρι μέσα Δεκεμβρίου. Άρα, για να δώσουμε τις δυνατότητε στις περιφέρειες να έχουν τους πόρους από τον νέο προπολογισμό, χρειαζόμαστε μια μεταβατική ρύθμιση. Και αυτό επειδή δεν μπορούμε να χάσουμε ένα-δύο χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε και την πράσινη συμφωνία. Θα πρέπει στην τρέχουσα περίοδο που περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία για την αλλαγή του κλίματος, για την προστασία του περιβάλλοντος, να συνεχίσουμε αν δεν έχουμε ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσει για το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο και για την πολιτική συνοχή για το γενικό κανονισμό. Θα πρέπει λοιπόν σε κάθε περίπτωση να τα προετοιμάσουμε αυτά. Και για το Κοινοβούλιο και για την Επιτροπή, αλλά και κυρίως για τις περιφέρειες θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μία επιπλέον ερώτηση να κάνω σε ό,τι αφορά αυτό το Ταμείο τη Μετάβασης. Γιατί είναι λίγο κάπως εξειδικευμένη αυτή η ερώτηση, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει να τη συζητήσουμε. Γιατί οι αρμοδιότητες δυστυχώς δεν είναι αποκλειστικά στα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό. Όταν ε, σε περιοχές λοιπόν ανθρακά ε, έχουμε βιομηχανίες οι οποίες είναι πολύ επιβαρυντικές ως το διδεξίδι του άνθρακα. Θεωρούμε ότι πρέπει να υποστηρίξουμε και θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις μεγάλες εταιρείες. Αυτή είναι η πρόταση την οποία καταθέσαμε, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να αλλάξουμε την ομοθεσία για τις επιδοτήσεις. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο η ομάδα μας ε, το έθεσε και στην πολιτική συνοχή να γίνουν λοιπόν επενδύσεις και στο Πράσινη Συμφωνία και στο Ταμείο Συνοχής και να μην υπολογιστούν στο ποσοστό χρέωσης. Να μην συνυπολογιστούν. Πώς ε, τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά το μέτρο αυτό. Ποια είναι η αποψή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κωνσταντ Κρέλε, η Επίτροπο τώρα έχει το λόγο για να απαντήσει. Σα ευχαριστώ πολύ και για να επανέλθω σε αυτά που είπα και προς τον κύριο Νοβακόφ. Προφανώς, νομίζω όλοι μας θέλουμε να ασκήσουμε πίεση στο Συμβούλιο προκειμένου να περάσει αυτή η τελική συμφωνία για το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό ζητάμε. Καταλαβαίνω φυσικά την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου. Να δούμε λοιπόν πώς θα αναπτύξουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία επεξεργαζόμαστε σε ό,τι αφορά τον κανονισμό, σε ό,τι αφορά την ρύθμιση. Γιατί ενδεχομένως η στρατηγική να λειτουργήσει και ξαφνικά να υπάρξει μια τελική συμφωνία σε ό,τι αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Λέτε και το παρατηρώ αυτό, αυτό ε, θα θέλαμε, αλλά δεν έχει συμβεί ως τώρα. Μπορεί όμως ακόμα να επιταχυνθεί ξαφνικά η διαδικασία και να ολοκληρωθεί. Δεδομένου λοιπόν των συνθήκων, πιστεύω ότι καλό θα ήταν να μην βρεθούμε χωρί τον απαραίτητο, τι απαραίτητε ρυθμίσει. Να είναι έτοιμε, δηλαδή. Ούτε να βρεθούμε σε μια κατάσταση που δεν θα είναι ενήμερα τα κράτη-μέλη και τα οργανωμένα τα κρατημέλη. Αυτά εννοούσα όταν ε, μιλούσα για μεταβατική περίοδος, περίοδο. Θα πρέπει να τα συζητήσουμε λοιπόν αυτά. Δεν πιστεύω ότι είναι επαρκέ στο πλαίσιο. Θα πρέπει να επισέλθουμε σε μεγαλύτερο βαθμό λεπτομερία. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται και στι επιτροπέ. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι η νομοθεσία, ο κανονισμό μάλλον, επί του οποίου έχουμε σημειώσει πρόοδο πριν τα Χριστούγεννα, δεν θα πρέπει να σταματήσει να υφίσταται. Αναφέρατε και καλά στοιχεία, τα επιπλέον χρήματα για παράδειγμα. Αυτό είναι παντού στο σχέδιο κανονισμού για το Ταμείο Δικής Μετάβασης. Το είχαμε υποσχεθεί άλλωστε, ότι θα ζητήσουμε, για... θα ζητήσουμε επιπλέον πόρους. Επιπλέον πόρους για τα καινούργια προβλήματα που ανακύπτουν. Αυτό αποτελεί λοιπόν τη βάση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε το 4,5 που ήδη είναι πιο πολλά από τα 4,8 που είχε απαιτήσει το Κοινοβούλιο τότε. Είναι λοιπόν επιπλέον χρήματα, επιπλέον πόροι. Θα δούμε λοιπόν τώρα συγκεκριμένα τι, τι, πώς θα δημορφωθούν αυτοί οι πόροι, αλλά επί της αρχής αναφέρεται αυτό το ζήτημα. Ένα από τα άλλα στοιχεία που αναφέρεται. Η νομοθεσία για τι κρατικέ επιδοτήσει στο μηχανισμό για το Ταμείο Δική Μετάβαση. Συμπεριλαμβάνεται αυτή η δυνατότητα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι βιομηχανικέ εταιρείε, το πώ θα τι βοηθήσουμε να κάνουν τη μετάβαση, ακόμα και αν είναι μεγάλε εταιρείε, όχι μόνο μικρομεσαίες δηλαδή επιχειρήσεις, προφανώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσει υποστηρίζονται και για την ποικιλομορφία της οικονομικής βάσης των περιφερειών αυτών, αλλά ακόμα και οι μεγάλες ε, Βιομηχανικέ εταιρείε μπορούν να αποτελέσουν αποδέκτες της βοήθειας αυτής. Το πώς όλα αυτά θα κατανεμηθούν προκειμένου να δοθεί καλύτερη και μεγαλύτερη επίοικια σε ό,τι αφορά τους κανόνες ε, κρατικής επιδότησης, εδώ θα πρέπει να κοιτάξουμε τους ίδιους τους κανόνες, γιατί το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε είναι ένα πλαίσιο το οποίο είναι περιορισμένο από την περιφερειακή πολιτική και από την πολιτική συνοχή. Αυτό που θα πρέπει να αποφύγουμε λοιπόν είναι να χρησιμοποιηθεί το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για να ανοίξουν εντελώς οι ρυθμίσεις της νομοθεσίας κρατικών επιτετήσεων χωρίς κανένα περιορισμό. Είναι περίπλοκο το θέμα και θα το κοιτάξουμε με την κυρία Φεστάγκερ για να δούμε πώς μπορούμε όλα αυτά να τα ρυθμίσουμε επακριβώς, αλλά σημαντικό είναι να έχουμε υπόψη μας ότι οι χώρες που μπορούν να πληρώσουν, να επιδοτήσουν τις μεγάλες εταιρείες, να μην καταλήξουν τελικά να εντείνουν τις ανισότητες σε σχέση με τις πιο φτωχές περιοχές. Αυτή είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Έχουμε ήδη κάποια περιθώρια για τη χαλάρωση των πολύ αυστηρών προτύπων και προδιαγραφών του προηγούμενου, της προηγούμενης νομοθεσίας. Αυτά περιλαμβάνονται στο μηχανισμό δίκαιης μετάβασης, αλλά για περαιτέρω χαλάρωση θα πρέπει να υπάρξει πιο ε, εκτενής συζήτηση. Προφανώς και με την μεγάλη συμμετοχή της Επιτρόπου Φιστάγκερ. Για να ξέρουμε τι ακριβώς κάνουμε. Μην καταλήξουμε τελικά για να λύσουμε ένα μικρό πρόβλημα, να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Για αυτό το golden rule, αυτό το, τη τομή. Ε, θα πρέπει να αναμνύουμε τις μεταρρυθμίσεις και τις αναθεωρήσεις το Φεβρουάριο. Κάτι που έχουμε συζητήσει όμως στο παρελθόν. Και κάτι το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε και να το σκεφτούμε. Γιατί ζητούμε μεγάλη συμμετοχή των ε, πόρων. Και κάποια κράτη-μέλη ενδεχομένω να χρησιμοποιήσουν την εθνική του συμμετοχή. Για αυτή τη μεγάλη, αυτή, την τεράστια αυτή αλλαγή που συνεπάγεται η Πράσινη Συμφωνία, και σε ό,τι αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και όλα αυτά που προβλέπει. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τι γίνεται και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να εξετάσει το θέμα αυτό και να το εξετάσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Τζεντιλόνι για να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να δημορφώσουμε αυτή τη χρήση τομή για το τι ε, θεωρεί η Ευρώπη στρατηγικές επενδύσεις και τι όχι. Φυσικά όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα συζητήσουμε επισταμένως αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει προηγουμένως μια μεγάλη προετοιμασία για να μην διακυβεύσουμε αυτά που έχουμε ήδη πετύχει. Ευχαριστώ πολύ. Για το Ρινιού, Στεφάν Πίσου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, όλοι μας θυμόμαστε τα λόγια που χρησιμοποιήσατε κατά τη διάρκεια της ακρόασής σας. Όλοι μας θυμόμαστε την ισχυρή δέσμευση, την αταλάντευτη προσήλωση που εκφράσατε, ε, διότι είπατε ότι θα δουλέψετε για να φέρετε απαντήσεις, για να δώσετε απαντήσεις σε όλους τους Ευρωπαίους, από όλες τις γωνιές της Ευρώπης, όπου και αν ζουν αυτοί. Όλοι θυμούνται ότι αναλάβατε τη δέσμευση, η πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ο Ευρωπαίος πολίτης στις κατατόπους περιφέρειες να ληφθεί υπόψη και έχουμε αυτό το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση και είναι η ευκαιρία να αποδείξουμε όλοι ότι εμείς και εμείς και εσείς καταλάβαμε το μήνυμα που μας στείλαν οι εκλογείς μας στις τελευταίες εκλογές. Μας είπαν ξεκάθαρα ότι θέλουν περισσότερη Ευρώπη, αλλά μια Ευρώπη που να υπηρετεί τους λαούς και τις διάφορες επικράτειες, τις διάφορες περιφέρειες, τα διάφορα εδάφη. Είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι το μήνυμα ελήφθη, αλλά θα πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να σταθούμε στο ύψο των περιστάσεων, έτσι ώστε καμία περιφέρεια που βρίσκεται σε ευπαθή κατάσταση, σε μειονεκτική κατάσταση, είτε στην υπηρετική Ευρώπη είτε στην νησιωτική Ευρώπη, να μην ε, μένει πίσω. Στα νησιά, για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε, συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα που μολύνουν, ενώ έχουμε τις ε, ε, αιωλικές πηγές ενέργειας, την ηλιακή ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές. Άρα πρέπει να παίξουμε αυτά τα χαρτιά, πρέπει να, να έρθουμε σε αυτό το ραντεβού, να μην χάσουμε αυτό το τρένο. Είναι απαραίτητο να κερδίσουμε αυτό το στοίχημα, να δράσουμε γρήγορα για να δείξουμε ότι δεν είναι οι καλές προθέσεις μόνο, αλλά ότι πραγματικά άλλαξαν τα πράγματα. Σήμερα, τώρα, έχουμε την ευκαιρία κάτι να κάνουμε και αυτό σας ζητώ τα κράτη-μέλη θα χρειαστεί να προσδιορίσουν τα ίδια ποιε είναι οι περιφέρειε που θα είναι επιλέξιμε για αυτό το μηχανισμό, για αυτό το Ταμείο τη Δίκαιης μετάβαση, Ωστόσο, όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εφιστήσουν την προσοχή όλων στι ε, περιφέρειε και περιοχέ, είτε υπηρετικέ, είτε νησιωτικέ, είτε εξόχω απόκεντρε, ότι πρέπει να σταθούμε δίπλα του, να επενδύσουμε για να πετύχουν αυτή, την πρόκληση τη δίκαιη μετά. Ευχαριστούμε τον Στέφαν ή Επίτροπος, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Στεφάν, για τα καλά σας λόγια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πράγματι, στην ακρόαση μου εδώ έδωσα κάποιες υποσχέσεις και θα κάνω τα πάντα για να τις πετύχω και να τις στηρίσω. Υποσχέθηκα ότι θα αγωνιστώ για μια δίκαιη μετάβαση, για μια μετάβαση όπου ο κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος, εκεί όπου είναι ο πιο έντονος, να κάνουμε τα πάντα να μετριαστεί, να μετριαστεί για να αντιμετωπίσουμε τους πιο σοβαρούς κινδύνους. Και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε με την πρόταση μας. Καταρχάς, προσθέσαμε αυτά τα κονδύλια πέρα και πάνω από τους φακέλους και την υφιστάμενη ε, χρηματοδότηση για τη συνοχή και τη γεωργία. Από εκεί και πέρα. Αφήσαμε ένα παράθυρο, ένα άνοιγμα. Όλοι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση. Και αυτό το φάκελο τον επιλέγουμε και τον κατανέμουμε, το χρηματοδοτικό φάκελο, κατά αναλογία με τον άμεσο αντίκτυπο, με τη σχετική σοβαρότητα των κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων της εκάστοτε περιφέρειας, ανάλογα με την απώλεια των θέσεων εργασίας στην εξορρυκτική ή ρηπογόνο βιομηχανία, η οποία θα οδεύσει προσκλήσιμο. Άρα έχουμε δείκτες τους οποίους μοιραζόμαστε, ανάλογα και με το ποσοστό των εκπομπών. Ε, ρήπων από βιομηχανικές πηγές σε σχέση με την προστιθέμενη αξία που κομίζει η ίδια ρηπογόνος βιομηχανία στην εκάστοτε περιοχή. Άρα προσθέσαμε οικονομικά κριτήρια, προσθέσαμε το δίκτυο της απασχόλησης, πόσες δουλειές εξαρτώνται από αυτή την ε, βιομηχανία και έτσι αυτά ε, τα χρησιμοποιήσαμε για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο της μετάβασης. Και θέλω να προσθέσω και ένα στοιχείο πολύ ενδιαφέρον για την πολιτική της συνοχής, τη σχετική ευημερία των κρατών, των χωρών, στο βαθμό που χρησιμοποιείται αυτή η έννοια της σχετικής ευημερίας, δηλαδή για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερο μια περιφέρεια ε, μιας φτωχής χώρας σε σχέση με μια περιφέρεια που έχει μεν ανάγκη αλλά βρίσκεται σε μια χώρα η οποία μπορεί να τη στηρίξει. Και βέβαια οι χώρε πρέπει να κάνουν επιλογή μετά, να επιλέξουν τι περιφέρειε και να υποβάλουν προτάσει. Αυτό είναι εναπόκειται στι χώρε και στην, ε, ε, ε στο εκάστοτε κράτο. Πρέπει δηλαδή να φτιαχτεί ένα σχέδιο και οι χώρες να μπορούν να καταρτήσουν ένα σχέδιο το οποίο να είναι συμβατό με το Εθνικό Σχέδιο για την Οικολογική Μετάβαση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια όρια, κάποια κατόφλια όντως για την αξιοποίηση του νέου ταμείου. Κάποια ανώτατα όρια. Το ταμείο θα πρέπει να προσθεθεί ε, στη δέσμευση και στα κονδύλια που έχουν τεθεί κατά μέρο και από το Εθνικό Ταμείο αλλά και από το Κοινωνικό Ταμείο και το Περιφερειακό Ταμείο της Ευρωπαϊκής γιατί είναι και εθνικό το πρόβλημα, έτσι είναι κοινό για όλους. Αυτή τη δομή, αυτή τη διάρθρωση προσπάθησαμε να σας παρουσιάσουμε και πιστεύω ότι καθησυχάζονται όλες οι ανησυχίες, μπορέσαμε να καλύψουμε τα ε, μεγαλύτερα θέματα, να ικανοποιήσουμε αυτά τα οποία μας παρουσιάσατε εσείς ως κόκκινες γραμμές. Βέβαια υπάρχουν κάποια όρια για ορισμένες χώρες εξαιρετικά φτωχές που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Πράγματι εκεί δεν μπορούμε να δώσουμε το μισό ταμείο σε αυτά, υπάρχουν και κάποια όρια για τις ε, πιστώσεις που τίθενται κατά μέρο ανάλογα με τα εθνικά κονδύλια τα περιφερειακά. 20% είναι αυτό το όριο για την επίλυση των προβλημάτων αυτών των ε, προβληματικών περιοχών. Ε, αυτές οι περιφέρειες αντιμετωπίζουν όντως σοβαρά προβλήματα, αλλά έχουν κι άλλα, όχι μόνο αυτό της διοικής μετάβασης. Είναι δύσκολη αυτή η άσκηση ισορροπίας, 20% δηλαδή μέγιστο όριο χρηματοδότησης από το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση. Στόχος είναι να πάμε πάρα πολύ γρήγορα, να προχωρήσουμε γρήγορα, να κλείσει το θέμα γρήγορα. γιατί ε, όλα αυτά σχετίζονται με συζητήσεις που έχουμε διεξάγει και στο παρελθόν. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει οριστική λύση. Καταλαβαίνω τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις κατανοώ. Δεν θα τις αμφισβητήσω, ούτε θα τις σχολιάσω. Αυτά που είπε ο Πρόεδρός σας δηλαδή. Όμως ε, δεν σημαίνει ότι με τη δίκαιη μετάβαση ε, θα έχουμε υποδεέστερες λύσεις και δεν σημαίνει το ότι ασκώντας πίεση τελικά θα πετύχουμε λιγότερα. Αλλά να μένουμε σε αυτό το τέλμα της ΑΕΝΑΙΣ διαπραγμάτευσης είναι κάπως προβληματικό και να έχουμε μεταβατικές λύσεις επάπειρων είναι όντως πρόβλημα πολλά, σχέδια, πολλά πράγματα που έχουν σχέση με τη μετάβαση, τη δίκαιη μετάβαση, συνδέονται με την ε, τρέχουσα λειτουργία της διαδικασίας. Οι περιφέρειες έχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες από εμάς. και εξαρτώνται ιδιαιτέρως από το κατά πόσο θα κερδιθεί το στίχημα της δίκαιης μετάβασης. Πρέπει δηλαδή ήδη από σήμερα να αρχίσουμε να δουλεύουμε με, βάση τις εμπειρίες και τα διδάγματα που έχουν αντλήσει αυτές οι περιφέρειες στο παρελθόν. Και όλα τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει πρέπει να τα αξιοποιήσουμε, πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό είναι το πιο ευεργετικό και το πιο δύσκολο. Να πάρει κανείς αναχείρας μια περιφέρεια και μάλιστα από μια φτωχή χώρα που δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικέ και να προσπαθήσει να βρει εναλλακτικέ. Ποιες είναι οι νέες προκλήσεις. Ποιες είναι οι νέες γραμμές προόδου. Δηλαδή ποια κατεύθυνση θα μπορούσε να ακολουθήσει αυτή η περιφέρεια για να έχει πρόοδο, για να ελαχιστοποιηθεί το εργασιακό και το κοινωνικό στόχο, ε, ε, κόστος αλλά και το ε, πρόβλημα σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητα. Ευχαριστώ για τους πρασίνους ο συνάδελφος Νίνας Ήκλας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την Επίτροπο που προσήλθε. Έχω ε, ε, ορισμένες ερωτήσεις σε σχέση με το Ταμείο Μετάβασης, όπως παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Νομίζω ότι εκπροσωπώ όλους εδώ και τις περιφέρειες όταν μιλώ για την χρηματοδότηση. Στην ουσία πολλαπλασιάζουμε την ε, ίδια την ε, χρηματοδότηση για τη μετάβαση αυτή και χρησιμοποιούμε και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων παράλληλα. Μιλάμε για 7,5 δις, άρα μιλάμε για μία αδύναμη ραχοκοκαλιά. Εσείς ε, προσβλέπετε σε μεγαλύτερη χρηματοδότηση για αυτό το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Υπάρχει δυνατότητα επαύξησης της χρηματοδότησης μέσω του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Η άλλη ερώτηση αφορά την συγχρηματοδότηση των διαρθρωτικών ταμείων. Αυτό είναι πολύ περίπλοκο ε, υπάρχει ένα θεωρητικό πλαίσιο εφαρμογής, αλλά δεν θα πρέπει να μεταφέρουμε ε, χρήματα από τη μία περιφέρεια στην άλλη. Δεν μπορούμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, να πούμε ότι α, αυτή η περιφέρεια είναι πιο σημαντική από την προηγούμενη και έτσι να μεταφέρουμε τα χρήματα από τη μία περιφέρεια στην άλλη. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία που θα είχαν ε, ήδη ενταχθεί σε αυτές τις ε, περιφέρειες. Ή μπορούμε να έχουμε περισσότερη, μεγαλύτερη χρηματοδότηση για το ε, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Πώς μπορεί δηλαδή να ε, διανεμηθεί αυτή η συγχρηματοδότηση ως προς την κλίδα κατανομής. Δεν υπάρχει ουσιαστική μεθοδολογία που να διέπει αυτή την κλίδα κατανομής. Γιατί δύο εκατομμύρια ε, δύο δις συγγνώμη, για την Πολωνία ή 900 εκατομμύρια για τη Γερμανία. Δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να μας επεξηγήσετε αυτή την κλίδα κατανομής για να κατανοήσουμε και τα αριθμητικά στοιχεία. Μπορείτε να μας δώσετε απαντήσεις και γραπτός. Και έπειτα αυτό το θέμα που έθιξε η Κωνσταντς των κρατικών επιδοτήσεων. Εδώ ακροβατούμε. Γιατί δεν θέλουμε να δούμε το εξής. Οι επιχειρήσεις που τα τελευταία χρόνια και δεκαετίες κατέστρεψαν το περιβάλλον και μας έφτασαν στην παρούσα κατάσταση όπου πρέπει να κάνουμε μία κατανομή χρημάτων για να απαλυνθούν τα αποτελέσματα της μόλυνσης του περιβάλλοντος, ότι αυτές οι επιχειρήσεις τώρα θα πρέπει να πάρουν επιπλέον χρήματα για να συνεχίσουν να καταστρέφουν το περιβάλλον. Είναι πολύ δύσκολο να το επεξηγήσουμε αυτό στους πολίτες. Όπως σας είπα, ε, στην ουσία βρισκόμαστε στο χείλος του γκρεμού γιατί δεν θα ήθελα να υπάρξει ε, απώλεια θέσεων εργασίας. Εντάξει, θέλουμε να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει κρατική επιδότηση για να υποστηρίξουμε απαρχαιωμένες μεθόδους και επιχειρήσεις που δεν έχουν θέση στο μέλλον. Πώς θα απομακρυνθούμε από το χείλος του γκρεμού. Και τα χρήματα αυτά να ε, δοθούν σε εργαζόμενους και όχι τους μετόχους. Ως προς την αιρεσιμότητα, αυτό που δεν κατανοώ στην πρότασή σας και ανοίγω μία παρένθεση για να πω ότι η πρόταση αυτή ήταν πολύ καλή ως προς τα κοινωνικά μέτρα και τον αποκλεισμό χρηματοδότησης για τα ορυκτά καύσιμα, αλλά δεν υπάρχει η σωστή ρεσιμότητα εδώ. Όταν δεν υπάρχει πλέον άνθρακας, τι θα προβλεφθεί για αυτές τις περιφέρειες. Θα υπάρχει ένα σχέδιο για το πώς μια συγκεκριμένη περιφέρεια μπορεί να απομακρυνθεί από τη χρήση άνθρακα. Γιατί μπορεί μια ε, περιφέρεια που να ζητήσει ε, που να ζητήσει τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Δίκαιη μετάβαση για να απομακρυνθεί από τον άνθρακα, αλλά στην ουσία δεν απομακρύνεται από τη χρήση άνθρακα, γιατί αυτό το Ταμείο δίκαιη Μετάβασης θα πρέπει να προβαίνει σε χρηματοδότηση όταν γίνεται ουσιαστική μετάβαση και απομάκρυνση από, τον, από τη χρήση άνθρακα. Ευχαριστούμε. Σας ε, υποβλήθηκε αυτή η συγκεκριμένη ερώτηση, η οποία θίγει ε, πολλές πτυχές ε, του ιδίου θέματος και θα θέλαμε μία απάντηση. Η Επίτροπος, ε, κύριε Νίκλας Νίνες, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις ερωτήσεις. Νομίζω ότι όταν αναφερθήκατε μάλλον η πρώτη σας ερώτηση σχετίζεται με τη χρηματοδότηση. Λέτε ότι το 7,5 ίσως να μην είναι επαρκές. 7,5. Οι συζητήσεις άρχισαν γιατί είπαμε ότι χρειαζόμαστε μία ευρωστότητα εκεί που δεν υπάρχουν χρήματα και θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον προϋπολογισμό πρωτίστως όχι μόνο ε, εξαιτίας της πίεσης από χώρες εκτός Ευρώπης που πιέζουν τις περιφέρειες και τις κοινωνίες της Ευρώπης. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε αντισταθμιστικά μέτρα, αλλά διότι ως Ευρωπαίοι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, μεγάλες προκλήσεις που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Είναι βέβαια πολύ δαπανήρη αυτή η λύση. Το πράσινο σύμφωνο είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο. Είχαμε προτείνει 4,8 το 2018 αρχικά και θεωρήσαμε ότι χρειαζόμαστε περαιτέρω χρηματοδότηση, γι' αυτό προτάθηκε το 7,5, δηλαδή φρέσκο χρήμα. Νομίζω ότι υπάρχει ενδυνάμει ζήτηση και αυτό το βλέπουμε όταν ε, αντιμετωπίζουμε τις επιμέρους καταστάσεις των περιφερειών. Μιλάμε λοιπόν για νέο χρήμα, αλλά θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφές. Η διάσταση αυτή του Πράσινου Συμφώνου δεν θα αφορά μόνο το δημόσιο κορβανά ή αυτά τα επιπρόσθετα χρήματα. Θα πρέπει να βρούμε και άλλες πηγές χρηματοδότησης για να συμμετάσχει και ο ιδιωτικός τομέας. Υπάρχει μεγάλη ρευστότητα στην αγορά η οποία αποζητά επενδύσεις Γι' αυτό εμείς θα πρέπει να διανοίξουμε ένα αυλάκι και να δείξουμε στην αγορά ε, τι επικερδή σχέδια και δυνατότητες υπάρχουν και αυτό μπορούμε να το δούμε και για τις ΜΜΕ, για τις θέσεις εργασίας και τις οικονομικές δραστηριότητες, παρά να μιλάμε για κερδοσκοπία. Αν είναι δυνατόν λοιπόν να έχουμε περισσότερα, ακόμα καλύτερα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα λογικό επίπεδο επενδύσεων, εάν λάβουμε υπόψη ότι μπορεί έτσι να εκκινήσουν και όλα τα άλλα στοιχεία τα οποία γνωρίζετε. Το EU Invest, αυτό το ταμείο, καθώς και η, χρηματοδότηση της ΕΤΕ και ούτω καθεξής. Αυτό το πακέτο είναι επαρκές. Είτε μιλάμε για 7,5 είτε μιλάμε για 200 δις. Βεβαίως τα 7,5 δις είναι το νέο χρήμα με στόχο τις περιφέρειες για να αντιμετωπίσουμε τις περιφερειακές πολιτικές και τις επενδυτικές πολιτικές των ε, περιφερειών, καθώς και τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο αυτών των περιφερειών. Πρόκειται για μία καθαρά περιφερειακή προσέγγιση. Όλα τα άλλα θα πρέπει να ενταχθούν στη, στα, στους σωστούς θύλακες χρηματοδότησης. Μιλάμε για, τον, για τον, την περιοχή 1. Αλλά μετά υπάρχουν και οι 2 και 3, EU Invest και μετά το μέσον συνδέοντας την Ευρώπη. Συγχρηματοδότηση τώρα. Αυτό είναι περιφερειακό πρόβλημα και είναι και το σημαντικότερο. Εμείς θεωρήσαμε ότι οι χώρες θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη διάσταση αυτού του ζητήματος. Οι χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα σε μία περιφέρεια δεν πρέπει να την αγνοήσουν. Θα πρέπει λοιπόν να επιληθούν αυτά τα ε, θέματα και κρατικά και διαπεριφερειακά, διότι το νέο αυτό χρήμα μπορεί να συνδυαστεί με ένα ελάχιστο 1,5 ευρώ ανά 1 ευρώ, αλλά μπορούμε να φτάσουμε και στην αναλογία 3 προς 1. Γι' αυτό ο συνολικός όγκος ε, διαφέρει. Μιλάμε για 30 ή 50 δις. Έχει σημασία κατά πόσο το κράτος μέλος θέλει να επιλύσει το εν λόγω ζήτημα. Εμείς λοιπόν έχουμε θέσει ένα όριο στη χρήση των ε, εθνικών χρηματοδοτήσεων. Υπάρχει το όριο του 20% για να απαντηθεί το ερώτημά σας. Δεν θα πρέπει να αποκλίνουμε από τα άλλα περιφερειακά ζητήματα. Στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε ζητήματα λεπτομερίας. Σημαντικά βέβαια. Τα ταμεία αυτά δεν αντισταθμίζουν τις ζημίες επιχειρήσεων. Όχι. Με τον μηχανισμό δίκαιης μετάβασης μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις που θέλουν να προβούν πραγματικά σε μία μετάβαση προς μία νέα τεχνολογία. Μπορούν να τύχουν υποστήριξης μέσα στα πλαίσια μίας χρηματοδότησης με το EU Invest, γιατί πρόκειται για μία ε, τραπεζική μετάβαση, η οποία μπορεί να τύχει υποστήριξης. Όπως ξέρετε δεν προβλέπεται από την νομοθεσία η κάλυψη της αρχής ορυπαίνουν πληρώνει. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες των ορυχείων θα έπρεπε να πληρώσουν για αυτό που προϋπήρχε. Αυτή ήταν η δική τους ευθύνη, είναι υπόλογη. Θα πρέπει όμως να, υπάρχουν, να υπάρχει χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που εργάστηκαν για 20-30 χρόνια ή και παραπάνω να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Για την απορρίπανση των ορυχείων, κάτι το οποίο δεν καλύπτεται εδώ. Εδώ καλύπτουμε τη μετάβαση μόνο, την επιχειρηματική μετάβαση, που χρησιμοποιούμε η απαρχαιωμένη τεχνολογία και πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες. Αυτός είναι και ο στόχος αυτής της υποστήριξης. Μετά αναφερθήκατε σε ορισμένα στοιχεία που άπτονται της αιρεσιμότητας και των πραγματικών επιπτώσεων αυτής της μετάβασης. Η αιρεσιμότητα σχετίζεται με το εξής. Για κάθε περιφέρεια χρειαζόσαστε ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο, το οποίο στη συνέχεια ε, οδηγεί στην σύμπραξη των περιφερειακών αρχών με τις εθνικές αρχές. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατότητα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για να οργανώσουμε ένα σχέδιο μετάβασης. Δηλαδή, έχουμε λύσει το θέμα ε, της μετάβασης, αλλά προς τα πού θα κινηθούμε. Αυτό το σχέδιο μετάβασης θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα εθνικά ε, ενεργειακά σχέδια και εθνικά σχέδια ως προς την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Θα ε, είναι σε επίπεδο ΝΑΤΣ 3, αλλά αυτή η μετάβαση θα πρέπει να διέπεται από μία συνοχή. Κάτι το οποίο δεν προανέφερα είναι το εξής. Είπατε, ε, δεν ξέρετε πως έχει αυτή η κλίδα κατανομής. Εμείς αρχίσαμε με τις περιφέρειες σε επίπεδο ΝΑΤΣ 3 και είδαμε ποιες είναι οι εκπομπές κατά κεφαλή. Ποιο είναι το επίπεδο εκπομπών ανακεφαλή. Μετά υποστηρίξαμε μάλλον υπολογίσαμε και τις εκπομπές θερμοκηπίου αναπεριφέρεια με βάση τα δεδομένα και των βιομηχανιών και μετά το κάναμε σε, επίπεδο, σε συνολικό επίπεδο βιομηχανιών με, ε, ε, με βάση και, την, ε, και, τον, και τις χιστολιθικές εξορίξεις και τα, τις πετρελαϊκές εξορίξεις και είδαμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Αυτό σχετίζεται με το ίμιση της απασχολησιμότητας, γιατί υπάρχει υψηλή απασχολησιμότητα τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη έκκληση άνθρακα, επίσης στις μονάδες λιγνίτη και στις ε, μονάδες εντατικής παραγωγής. Έχουμε συγκεκριμένους δείκτες και φτάσαμε σε έναν μαθηματικό τύπο για κάθε κράτος μέλος. Μετά προβήκαμε σε μία οριοθέτηση, διότι φιλτράραμε όλα αυτά τα στοιχεία, είδαμε την σχετική ευημερία της χώρας, για να μην ε, προβούμε σε υπερβάσεις, σε σχέση με τις χώρες που έχουν μεγάλη χρηματοδότηση, χρησιμοποίησαμε την φόρμουλα του Βερολίνου και μετά θέσαμε ορισμένα όρια για το πόσο χρήματα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε κράτος μέλος. Και έτσι φτάσαμε σε ένα ανώτατο όριο. Αυτός, ε, αυτός είναι ο συνδυασμός τη, του μαθηματικού τύπου που βλέπετε στο παράρτημα 1. Αυτό ακριβώς κάναμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Από πλευρά του ΕΛΚ το λόγο έχει η κυρία Ντονατό. Ευχαριστώ πολύ και θα μιλήσω τελικά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επίτροπο για την διαθεσιμότητά της που βρίσκεται εδώ και για διεξοδικές απαντήσεις που έδωσε μέχρι τούδες του συναδέλφους. Θα ήθελα να πω ότι από τις απαντήσεις σας έχω λάβει αρκετές διευκρινήσεις, διευκρινιστικές επεξηγήσεις. Θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι την ανάγκη της επιτάχυνσης των ορισμών των κανονισμών ως προς τα διαρθρωτικά ταμεία και του κοινού κανόνες ε, ιδιαίτερα σε σχέση με το νέο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και θεωρώ όπως προελέχθη ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας μεταβατικός κανονισμός αλλά οι καθυστερήσεις που θα υπάρξουν δεν θα πρέπει να υπερβούν το έτος γιατί η έλλειψη συμφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν πολύ αρνητικό μήνυμα για τους πολίτες και θα αποδυνάμωνε την εργασία μας για τη συνοχή. Υπάρχει ανάγκη να είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές συνοχής, γιατί μιλάμε για χορήγηση πιστώσεων, για χρηματοδοτήσεις, αλλά ε, ακριβώς επειδή γίνονται πολλαπλές χρηματοδοτήσεις, στη συνέχεια είναι δύσκολο να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη χρηματοδότηση ορισμένες περιφέρειες της Ευρώπης. Για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο, θα πρέπει στη νομοθετική σας εργασία και τη δική μας νομοθετική εργασία, να ληφθούν υπόψη όλες οι πολιτικές ομάδες που εκπροσωπούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Με βάση την δημοκρατική αντιπροσωπευτικότητα και θα προέτρεπα το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τις απαιτήσει όλων των κρατών μελών, όπως και εσείς υπογραμμίσατε, τις χώρες που έχουν ανάγκη από πολιτική συνοχής, δηλαδή που γνωρίζουν μεγάλες καθυστερήσεις σε σχέση με άλλες περιφέρειες. Θα πρέπει λοιπόν να προβούμε σε μία μεταρρύθμιση των κρατικών επιδοτήσεων και αυτό για να μπορέσουμε να διευρύνουμε το πλαίσιο χρηματοδότησης υπέρ της ε, εδαφικής συνοχής. Μεγαλύτερη λοιπόν ευελιξία και μεγαλύτερο άνοιγμα των κρατικών ε, επιδοτήσεων τη στιγμή που δεν υποστηρίζουν τις ιδιαίτερα αναπτυγμένες περιφέρειες και επιχειρηματικές οντότητες, αλλά όταν πρόκειται για την ανάπτυξη των πλέον απομακρυσμένων και μειονεκτουσών περιφερειών. Όπως είπατε και το εκτίμησα ιδιαίτερα, μας ενδιαφέρει και ο εξυγχρονισμός του ε, Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για να ληφθεί υπόψη και ο χρυσός κανόνας και οι χώρες που δεν έχουν μεγάλες δυνατότητες χρηματοδότησης να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Τέλος, θα ήθελα να υποβάλω μία ερώτηση σε σχέση με την εφαρμογή του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Γιατί θεωρούμε ότι αυτή η εφαρμογή θα πρέπει να είναι η ευρύτερη δυνατή. για να μην πάνε αυτά τα χρήματα σε αυτούς που είναι ε, καθαροί εισφορείς ή σε περιφέρειες που χαίρουν άκρας υγείας. θα πρέπει να πρόκειται για περιφέρειες ε, που προβάλλουν καθαρότερες πηγές ενέργειας, ενέργειας όχι δηλαδή ε, ανθρακογόνες. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι οδικές μεταφορές ε, ρηπαίνουν. Δηλαδή πάλι έχουμε ε, εκπομπές θερμοκηπίου. Θεωρώ λοιπόν ότι η μετάβαση από τις οδικές μεταφορές στις σιδηροδρομικές θα ήταν κάτι το πολύ θετικό. Αυτό αφορά και τις ε, απαρχαιωμένες μονάδες που παράγουν χάλιβα, τις μεγάλες χαλιβουργίες που ρηπαίνουν το περιβάλλον. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που στην ουσία οδηγούν στην μείωση ρηπογόνων εκπομπών. γιατί έτσι θα μειωθούν οι εκπομπές θερμοκηπίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αναμένω τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ, συνάδελφε, και τον λόγο έχει η Επιτροπή για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Φραντσέσκα Ντονάτο. Σημειώνω τα μηνύματα τα οποία μας αναφέρετε. Ανέφερα ακριβώς και εδώ πιστεύω ότι υπάρχει σύγκληση και είναι σημαντικό να έχει ολοκληρωθεί ο κανονισμός και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να έχει οριστεί. Δεν θέλω ο μεταβατικό μηχανισμό, εάν και εφόσον αποφασιστεί και πάντα θα αποτελέσει τη δεύτερη καλύτερη λύση, γιατί προφανώ και θα δημιουργεί αστάθεια, αντί λοιπόν να ασκήσει η πίεση, να δώσει μια ανακούφιση, ανακούφιση και να καθυστερήσει περαιτέρω την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε λοιπόν την πίεση και να δαπανίσουμε ενέργεια όχι προ την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, αλλά προ άλλο σκοπό. Συμφωνώ από αυτού. Κάνατε διάφορα σχόλια. Σχόλια τα οποία ήδη έχουν αντιμετωπιστεί και είναι σημαντικό οι πιο ασθενείς χώρες να μην εμποδιστούν λόγω αδυναμίας χρήσης των δικών τους πόρους, του εθνικού σκέλους της χρηματοδότησης. Θα δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Όπως ξέρετε, στην πολιτική συνοχή έχουμε ήδη εισάγει διαφορετικά επίπεδα ζήτησης σε ό,τι αφορά τους εθνικούς πόρους, ανάλογα και με το οικονομικό επίπεδο των περιοχών και των χωρών. Εδώ επιδεικνύουμε μεγάλη προσοχή, το εξετάζουμε πολύ προσεκτικά. Αναφερθήκατε στη συνέχεια και κάνετε πολλά σχόλια τα οποία είναι πολύ επίκαιρα σε ό,τι αφορά την χρήση γενικά της πολιτικής συνοχής. Εδώ θα ήθελα να τονίσω κάτι. Σε κάποιες περιπτώσεις, στον κανονικό διάλογο, ο κόσμος λέει, και εγώ προσπαθώ πάντα να το διορθώσω, ότι υπάρχει μια παλιά πολιτική, η πολιτική συνεχή και ότι υπάρχει και η καινούργια πολιτική, οι καινούργιες πολιτικές. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνούμε με τέτοιου είδους δηλώσεις, γιατί στην πολιτική συνοχή έχουμε κάποια εργαλεία και έχουμε επισημάνει την πολιτική συνοχή. Όταν μιλάμε για ασθενείς περιοχές, όταν μιλάμε για συστήματα μεταφορών, να γίνονται μεταφορές αυτές ανάλογα με τις απαιτήσει του περιβάλλοντος. Δεν μπορούμε δηλαδή να βασιστούμε σε παλιές τεχνολογίες που θα έχουν και μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Πρέπει να πρασινίσει λοιπόν η περιφερειακή πολιτική και όλα τα εργαλεία της περιφερειακής πολιτικής και γι' αυτό το λόγο έχουμε ε, συγκεκριμένα αναθέσει τους πόρους αυτούς προς την κατεύθυνση αυτή για να υπάρχουν οι ανάλογες επενδύσεις και μάλιστα με το βλέμμα προς το μέλλον, όχι στο παρελθόν λαμβάνοντας υπόψη και τους περιβαλλοντικούς κανόνες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το στοιχείο αυτό. Ύστερα, μιλήσατε για το σύστημα μεταφορών, για τις βιομηχανίες στο σύνολο τους. Ο μηχανισμός αυτός μετάβασης είναι κάτι το επιπλέον για να αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε απαντήσεις στην τραγική αυτή εικόνα την οποία έχουν σε κάποιες περιπτώσεις οι περιφέρειες ε, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της μετάβασης. Όταν τα προβλήματα λοιπόν είναι ιδιαίτερα σοβαρά, υπάρχει αυτή η επιπλέον βοήθεια. Σε ό,τι αφορά το γενικό σύστημα μεταφορών τώρα, σε ό,τι αφορά τις μονώσεις στις κατοικίες για νέες ε, νέου τρόπου μετάβαση βιομηχανιών κτλ. Έχουμε όλα τα εργαλεία στη διάθεσή μα και να μην ξεχνάτε ότι μαζί με το μηχανισμό δίκαιη μετάβαση έχουμε και ένα-τρει ε, επενδύσει που έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το επεξεργάζονται αυτό οι συνάδελφοι τη Επιτροπής, γιατί η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί μια επανάσταση στον τρόπο παραγωγής, τίποτα δεν θα μείνει όπως πριν. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να κάνουν μαζικές επενδύσεις στον τρόπο παραγωγής τους, στη βελτίωση των τεχνολογιών τους για να καταστούμε παγκόσμιοι ηγέτες σε ό,τι αφορά τα... τις τεχνολογίες αυτές. Αυτό είναι το μέλλον. Αλλά εδώ δεν μπορούμε να στρεχτούμε αποκλειστικά και μόνο στο μηχανισμό δικής μετάβασης ή μόνο στον ευρωπαϊκό προπολογισμό, γιατί όλο το σύστημα θα πρέπει να δώσει απαντήσεις στις καινούργιες αυτές ανάγκες. Και εδώ πιστεύω ότι έχετε απόλυτο δίκιο, ανοίγοντα και τις άλλες διαστάσεις. Αλλά ασφαλώς αυτό που συνεπάγεται το στοιχείο αυτό είναι ότι όλος ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να στραφεί προς την κατεύθυνση αυτή και όχι να περιοριστούμε στα 7,5 δις. Είναι μεγάλο το ποσό, αλλά δεν μπορεί να επιλύσει όλα τα προβλήματα Χρειάζεται λοιπόν επιπλέον βοήθεια για να αντιμετωπιστούν τα πολύ σοβαρά και συγκεκριμένα ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής φύσεως που αντιμετωπίζουν κάποιες περιοχές. Αυτά ισχύουν λοιπόν. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Για τους ΕΣΥΑΡ, το λόγο έχει Ραφαήλ Φικό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω την Επίτροπο με χαρά την άκουσα και είχα παρευρεθεί και στην ακρόασή της και εκτίμησα τις ενδυνάμει αρμοδιότητές της μέσα στα πλαίσια του πολυσχηδούς αυτού τομέα που μας απασχολεί. Θα πρέπει να λάβουμε όμως υπόψη ότι όλα όσα προελέχθησαν σε σχέση με το νέο πράσινο σύμφωνο δεν μας βρίσκουν, μας βρίσκουν όλους ε, θεωρητικά σύμφωνους. Όσοι καταψήφισαν ε, δεν ε, αντιτίθενται στο περιεχόμενο, αλλά διότι στις συζητήσεις διείδαν μία ανικανότητα στο να τεθεί σε εφαρμογή αυτό το πλαίσιο. Δεν είμαι επικριτικός. Ελπίζω η παρούσα Επιτροπή να μπορέσει να δώσει μία νέα όθηση στο ολοζήτημα και αυτό έναντι του Συμβουλίου. Αλλά ποια είναι τα σημεία που θα πρέπει να υπογραμμιστούν για να δούμε εάν υπάρχει κάποια τροχοπέδη κατά αυτή την περίοδο. Η πρώτη ε, συνιστόσα που αφορά το ε, ταμείο αυτό δίκαιης μετάβασης αφορά κάτι το οποίο μπορεί να αμφισβητηθεί. Δηλαδή πώς η Ιταλία μπορεί να λάβει μόνο 364 εκατομμύρια για όλες τις ε, ανθρακοβόρες επιχειρήσεις και τη στιγμή που υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που θα κλείσουν. Αυτό είναι ιδιαίτερα άδικο και ετεροβαρές σε σχέση με τις επιλογές σας. Όταν μιλάμε για την πολιτική συνοχής, εσείς αναφερθήκατε στην ανάγκη της συγχρηματοδότησης. Δηλαδή μιλάμε για μία μονάδα που δεν χρησιμοποιεί μόνο ευρωπαϊκούς πόρους. Όταν γίνεται λόγος για σύμφωνο σταθερότητας, εγώ θα το ενέτασα σε αυτό το σκεπτικό. Γιατί φοβάμαι ότι πρώτα μιλάμε για το Ταμείο ε, Δίκαιης Μετάβασης, μετά θα μιλήσουμε για το ε, Πράσινο Σύμφωνο και μετά θα μιλήσουμε για το σύμφωνο σταθερότητας. Δηλαδή γίνεται μία κακή ιεράρχηση και στην ουσία η απότερη βλάβη θα αφορά το Ταμείο Συνοχής, την πολιτική συνοχής, διότι το τελευταίο εξάμεινο υποβλήθηκε μια πρόταση που κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή η πολιτική συνοχής πολύ δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Επειδή λοιπόν προκύπτουν δυσκολίες, υπάρχει ο φόβος ότι στο τέλος θα βλαφθεί η πολιτική συνοχής, διότι ήδη έχουν γίνει καθυστερήσεις εξ αρχής και γι' αυτό μιλώ, για αυτή τη μεγάλη ανησυχία και θεωρώ ότι η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκφράσουν αυτές τις ανησυχίες, διότι βαθμιαία φτάνουμε και στην αναπομπή ε, του προγραμματισμού αυτού και έτσι φτάνουμε λαμβάνουμε γνώση του γεγονότος ότι επί επιπροσθέτως μειώνονται τα κονδύλια προς την πολιτική συνοχή. Αυτός, αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία, γιατί όσο περισσότεροι και να είναι οι πόροι, το ε, νέο πράσινο σύμφωνο δεν μας οδηγεί σε μια μεγάλη σιγουριά. Μιλάμε για χίλια δις, αλλά δεν έχουμε καμία ε, σιγουριά για την πρόελευση αυτών των πόρων. Και δεν θα ήθελα μέσα σε όλα αυτά να βλαφθεί η πολιτική συνοχής, να καταβάλει ένα τόσο υψηλό τίμημα. Γι' αυτό θα πρέπει να διασαφηνίσουμε ορισμένα βασικά ζητήματα και ελπίζω έτσι να μην υπάρξει καμία βλάβη και να μην επικρατήσουν άλλες πολιτικές έναντι της πολιτικής συνοχής. Δηλαδή να μην καπελωθεί αν θέλετε η πολιτική συνοχής από άλλες πολιτικές και μέσα. γιατί όπως ξέρετε η κάθε πολιτική έχει συγκεκριμένες συνιστώσεις. Ελπίζω λοιπόν να υποστηρίξετε αυτή τη δράση υπέρ της πολιτικής συνοχής πρωτίστως. Σας ευχαριστώ πολύ Ραφαέλ και το λόγο έχει η Επιτροπός. Ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι επισημάνονται πολλές ανησυχίες. Γιατί είμαι υπέρ τη ε, Πράσινη Συμφωνία, Γιατί νομίζω ότι πολύ απλά δεν έχουμε εναλλακτική. Θα πρέπει να το πετύχουμε, θα πρέπει να πετύχουμε κάτι. Και αντιλαμβάνομαι, όπω και όλοι μα άλλωστε, ότι υπάρχει αυτή η εξωτερική διάσταση. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Το οποίο και το κάναμε. Γι' αυτό λοιπόν είμαι υπέρ μεν αλλά θέλω να τοποθετηθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην ημερήσια διάταξή μας, προκειμένου αυτή η θετική εξέλιξη να μην καταλήξει να έχει αρνητικά προβλήματα τελικά. Γιατί η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ε, θέρμανση του πλανήτη και στα αέρια του θερμοκηπίου είναι 9%, αλλά η παρουσία μας, η εμπορική, σε παγκόσμιο επίπεδο είναι εξαιρετικά ισχυρή. Όπως και αν τα μετρήσουμε τα πράγματα, εξακολουθούμε να είμαστε η μεγαλύτερη τέτοια εμπορική δύναμη. Άρα η εξωτερική διάσταση της Πράσινης Συμφωνίας θα πρέπει προφανώς να αναλυθεί μαζί με την διπλωματική μας ικανότητα προκειμένου στο παγκόσμιο προσκήνιο να διαδραματίσουμε το ρόλο που μας αναλογεί για τον νέο τρόπο παραγωγής. Αλλά πραγματικά δεν πρέπει να καταρρεύσει ο πλανήτης. Το βλέπουμε να συμβαίνει καθημερινά. Είναι αναπόφευκτο. Και έχουμε το μερίδιο της ευθύνη μας. Και πραγματικά όλοι από εμά περιμένουμε και ο κόσμος στον δρόμο καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει τη διαδικασία αυτή για το Ταμείο Δικής Μετάβασης. Δημιουργούμε πιο πολλά εργαλεία για να αποφύγουμε τον περίπλοκο αυτό χαρακτήρα και δύο στοιχεία θεωρώ ότι θα πρέπει να τονίσουμε. Το ένα είναι ότι αυτός ο μηχανισμός δίκαιης μετάβασης αφενός κατοχυρώνεται στο πολίτης δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να τοποθετηθεί στο επίκεντρο του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου και από την άλλη στο Ταμείο περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν το γεγονός είναι που θα χρησιμοποιηθεί για να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα σε κάποιες περιοχές. Αλλά προκειμένου να λειτουργήσει σωστά ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Και πάλι λοιπόν, προφανώς ανακύπτει το πολιτικό ερώτημα. Όλοι σας φαντάζομαι. Είσαστε άλλωστε και πολιτικοί. Θα πρέπει να καταβάλουμε μια προσπάθεια λοιπόν για να περιορίσουμε την επίπτωση και τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Μιλάμε για το 1% του συνολικού πλούτου. Μπορούμε όμως σε αυτό το επίπεδο ενοποίησης να έχουμε έναν σε εισαγωγικά ομοσπονδιακό κοινό προϋπολογισμό 1% του πλούτου μας. Σε καμία τέτοια περιοχή με πολλές χώρες δεν μπορεί. Και εδώ κάνετε για παράδειγμα έναν, ε, μια σύγκριση με τον προπολογισμό της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ε, της, ε, των Η Γερμανία θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Η Ελβετία θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα χωρίς ομοσπονδιακό προπολογισμό. Μιλάμε για κάποια ελάχιστα επίπεδα τα οποία χρειάζονται για να σταθεροποιήσουν τον προπολογισμό. Και προφανώ η συζήτηση είναι πάρα πολύ εκτενή. Αλλά δεν συζητάμε τι γίνεται με την ευρωπαϊκή συνεισφορά του 99% του κοινού πλούτου. Και εδώ ε, μιλάμε για μεγαλύτερα ποσά, γιατί αφορά όλους μας αυτό, από κοινού. Θα πρέπει να δείξουμε λοιπόν στους πολίτες τι κάνουμε με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί πολλοί θεωρούν ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι απλά δαπάνες. Τι θα γινόταν, πού θα είμαστε, πού θα ήταν όλες αυτές οι χώρες και περιοχές που βρίσκονται εδώ πέρα και αντιπροσωπεύονται εδώ πέρα, αν δεν υπήρχε πολιτική συνοχή. Θα πρέπει να δείξουμε λοιπόν στους πολίτες και να πούμε στους πολίτες σοβαρούς πολιτικούς τι συμβαίνει και να εξηγήσουμε λοιπόν ακριβώς τι συμβαίνει, όχι απλά να περιοριστούμε σε γενικότητες. Γιατί πολύ απλά υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των περιφυγών που έχουν διαφορετικό επίπεδο και δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν προκειμένου λοιπόν να καταστεί αποδεκτός ο ανταγωνισμός. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει η πολιτική συνοχή και πραγματικά υπάρχουν κάποια βασικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επανέλθουν στην πολιτική συζήτηση. Έχουμε λοιπόν την επιλογή αυτή. Είναι να επικεντρωθούμε μόνο σε φτωχέ χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα μετάβασης σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές αλλά εδώ θεωρώ ότι οι πιο πλούσιες χώρες δεν θα καλύπτονταν από τον μηχανισμό μετάβασης. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε το εξή, να δώσουμε ευκαιρία σε όλα τα διάφορα κράτη-μέλη να έχουν πρόσβαση. Η Ιταλία, είπατε, ε, με τα μεγαλύτερα εργοστάσια χάλευα, αλλά με κατακεφαλήν ΑΕΠ που επιτρέπει τη χρήση και των δικών της πόρων για να επιδοτήσει τις βιομηχανίες της. Αυτό εννοείται με το στοιχείο σχετικής ευημερία. Αν συγκρίνουμε την Ιταλία με την Πολωνία, για παράδειγμα, κατά πάσα πιθανότητα, αν υπάρχουν πολύ αυστηρά κριτήρια, θα έπρεπε να υπάρξει ένα ταμείο για την Τσεχία, την Πολωνία, την Ρουμανία και όλες οι υπόλοιπε χώρες θα ήταν απούσες. Αυτό δεν το επιλέξαμε ω σύστημα. Προφανώ χρειάζεται μια εξισορρόπηση. Δεν λέω ότι είναι τέλειο το σύστημα. Σε εσά επαφίεται πλέον να τσεκάρετε τον κανονισμό, να συζητήσετε το μαθηματικό τύπο που χρησιμοποιείτε και να τον τροποποιήσετε. Έχει πιο πολύ νόημα όμω και οι χώρε που, όπω η Γερμανία, θεωρούνται και είναι καθαροί εισφορεί, επίση να ωφεληθούν στι πιο φτωχέ περιοχέ τους να έχουν και αυτές κάποια υποστήριξη. Αλλά αυτή η υποστήριξη κάπως να προσαρμοστεί και στο συνολικό πλούτο της χώρας, προκειμένου να συνυπολογιστεί η ικανότητα επίλυσης των δικών της προβλημάτων. Τίποτα δεν είναι τέλειο. Προφανώς πρόκειται για μια ισορροπία, την οποία προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να την προτείνουμε. Αλλά η επιλογή ήταν αυτή, προκειμένου να μην αποκλειστεί κανείς, να μείνει κανείς απ' έξω. Αλλά και στην Ιταλία, την 7η μεγαλύτερη οικονομία, υπάρχουν προβλήματα. Και θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη προς τις τοπικές τέτοιε εταιρείε. Τέτοιου είδους λύσεις ποτέ δεν είναι απόλυτα σωστές και άμεμπτες, αλλά αυτή είναι η καλύτερη δυνατή λύση που σκεφτήκαμε και σε σας επαφή ήταν τα εξετάστα λεφτά και έφυγε ο Νίκολας αλλά νομίζω ότι κατά πάσα πιθανότητα έκανε ένα λάθος όταν του είπα. Όταν κάναμε την πρώτη ανάλυση για τις περιφερειές και τις περιφερειές που ήταν πάνω από ή κάτω από το μέσο όρο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοιτάξαμε το ΝΑΤΣ 2 και τώρα όταν κάναμε την ε, εκτίμηση ήταν μέσα στο επίπεδο ΝΑΤΣ 3, σε πιο α, λεπτομερές επίπεδο, πιο μικρό επίπεδο. Μάλλον ε, λάθος έκανα εκείνη την ώρα. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες σας. Εγώ το βλέπω και από την άλλη πλευρά. Πρέπει να ολοκληρωθεί η ατζέντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ας συνεργαστούμε λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τα διάφορα στοιχεία. Αλλά προφανώς ε, είναι μία επιλογή. Μία επιλογή μεταξύ τη ανάγκης ε, υποστήριξη και τη ικανότητα των κρατών μελών να επιλύουν τα δικά του προβλήματα. Χρειάζεται λοιπόν να ε, δοθεί βοήθεια γιατί σε κάποιε περιπτώσει αυτέ οι περιφερειακέ ε, εταιρείε δεν είναι τόσο και οργανώσει δεν είναι τόσο πλούσιες όπω η χώρα του. Είμαστε λοιπόν εδώ όλοι μαζί για να σκεφτούμε ποια είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Γιατί όλοι μαζί είμαστε πιο ισχυροί από ό,τι καθένα μόνο του. Σα ευχαριστώ για τι πολύ ολοκληρωμένε απαντήσει σας. Για την ΚΟΕ, Μαρτίνα Μίτσελ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Επίτροπε. Και από δική μα πλευρά σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και καλή χρονιά. Και θα χρειαστεί προφανώς ε, μεγάλη υπομονή και επιμονή σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή. Θα σα υποστηρίζουμε. Υποστηρίζω ιδιαίτερα σε αυτά που είπατε για το θέμα του ότι δεν μπορούμε να τα πετύχουμε όλα και να τα βάλουμε όλα μέσα σε ένα πρόγραμμα. Χρειαζόμαστε διαφορετικά εργαλεία για μια πολιτική συνοχή. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε προς όλες τις πλευρές. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί Γι' αυτό λοιπόν μία ερώτηση να κάνω σε ό,τι αφορά τη δική μετάβαση. Εξ κατάλαβα, πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο κυρίω θα επικεντρωθεί στην αποχώρηση από τον άνθρακα. Τι θα κάνετε λοιπόν για να μην γίνει ένα πηγάδι χωρίς πάτο το θέμα αυτό. σε ό,τι αφορά την ε, ε, περιβαλλοντική επιβάρυνση. σε ό,τι είπατε για την επικεντρωσή σε κάποιες περιφέρειες κτλ. Θα επικεντρωθείτε μόνο στο θέμα αυτό ή θα κοιτάξετε και άλλα θέματα. Δεύτερη ερώτηση. Το ταμείο αυτό, εκτός όσων καταλαβαίνουμε, ουσιαστικά θέλει να βοηθήσει τον πολίτη τον εργαζόμενο, ο οποίος αισθάνεται ότι απειλείται από την απαχώρηση από τον άνθρακα ή και τις βιομηχανίες που στρέφονται προς ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Πώς θα τονίσετε λοιπόν το στοιχείο αυτό, προκειμένου να μην καταλήξει να είναι ένα πρόγραμμα επενδύσεων για τους μεγάλους ομίλους, για τις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες, αυτό θα ήταν ε, φυσικά λάθος και το είπατε ότι δεν είναι αυτό ο σκοπό σας, αλλά έχετε συγκεκριμένες ε, προτάσεις και σκέψεις για το πώς θα τονίσετε και την κοινωνική πτυχή, πώς θα βάλετε στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τον πολίτη. Τελευταία ερώτηση για το υποχρεωτικό, την υποχρεωτική ε, συνεισφορά των κρατών μελών για τον στόχο για την πράσινη Ευρώπη. Τι θα γίνει με το στοιχείο αυτό. Merci beaucoup, Ευχαριστώ Μαρτίνα. Κυρία Πίτροπε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας απαντούσα λέγοντας ότι ναι, απευθύνεται στις περιφέρειες. Προορίζεται για τις περιφέρειες, όχι όμως μόνο ε, για τις περιφέρειες που εξαρτώνται από το σχιστολιθικό αέριο, από το λιγνίτη, από τον άνθρακα. Όχι μόνο για αυτές. Απευθύνεται και στις ε, περιφέρειες όπου έχουμε βιομηχανία υψηλής εντάσεως εργασίας, όπου έχουμε υψηλή δηλαδή ε, ρηπογόνο δραστηριότητα και πρέπει να βοηθηθούν να κάνουν τη μετάβαση. Δεν μιλούμε μόνο για τον άνθρακα και την εξόριξη, είναι και οι βιομηχανίες οι εξαιρετικά ρηπογόνες, οι περιφέρειες όπου υπάρχουν τέτοιες θεωρήσαμε ότι δεν θα είχε νόημα να έχουμε ένα εργαλείο απόν περιμένοντας τα ανθρακοριχεία να κλείσουν ή τις βιομηχανίες να κλείσουν και στη συνέχεια να φτιάξουμε ένα εργαλείο για να στηρίξουμε τον κόσμο. Εάν ξέρουμε ότι υπάρχει συγκεκριμένη βιομηχανία που χρησιμοποιεί απαξιωμένη τεχνολογία και που χρειάζεται τη μετάβαση πρωτού κλείσει και χωρίς να κλείσει, τότε πρέπει να είμαστε παρόντες για να στηρίξουμε αυτή τη μετάβαση, για να μην σκοτώσουμε δηλαδή όλες τις δουλειές τις διαθέσιμες και να βρούμε λύσεις. Είναι βασικό συλλογισμός αυτός. Ε, αυτό είναι το σκεπτικό μας. Και είπατε και κάτι πολύ σημαντικό αν απλά κάνουμε διάχυση των χρημάτων ή αν θα επικεντρωθούμε στις κρίσιμες περιφέρειες. Απαντώ λέγοντας το δεύτερο. Πρέπει να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στις κρίσιμες σημασίας περιφέρειες. Βέβαια, είναι αρμοδιότητα του κράτους μέλους να μας προτείνει σε ποια περιφέρεια θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας. Αυτό πρέπει να γίνεται σε στενό διάλογο μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, σε σχέση και με το εξάμεινο, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, θα αναδείξουμε τους τομείς και τις περιοχές όπου περιμένουμε τη χώρα να λύσει τα προβλήματα. Άρα θα υπάρξει διάλογος για τα θέματα αυτά. και θέλουμε οι επιλεγήσεις περιοφέρειες και περιοχές όχι μόνο να είναι ιδιαίτερα εξαρτημένες από αυτές τις δραστηριότητες, αλλά να είναι και οι πιο φτωχές, να είναι και εκεί όπου είναι πιο δύσκολο να βρεθούν εναλλακτικέ. Αυτές τις περιφέρειες θέλουμε να, με αυτές θέλουμε να ασχοληθούμε και γι' αυτό επισκέπτομαι τέτοιες περιφέρειες στην Πολωνία, θα πάω και στην Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία, ήδη είχα πάει στην Ελλάδα στο παρελθόν. Έχω ήδη πάει. Και την επόμενη φορά που θα πάω, κατά πάσα πιθανότητα θα πάω στη Δυτική Μακεδονία, είναι οι κρίσιμε περιφερειές που έχουν οπισθοχωρήσει, που δεν έχουν πολλέ εναλλακτικέ και που εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο, αν όχι σε απόλυτο βαθμό, από αυτέ τι δραστηριότητε. Επομένω, με τη σταδιακή εξάλληψη αυτών των οικονομικών δραστηριοτήτων, τίθεται το μεγάλο ερώτημα τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πού θα δουλέψουν, ποια άλλη οικονομική δραστηριότητα θα αναλάβουν. Γι' αυτό λοιπόν Πρέπει να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας σε αυτές τις περιφέρειες συγκεκριμένα και δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε λίγα λεφτά σε πάρα πολλά διαφορετικά ε, πράγματα διάσπαρτα για να υπάρχει μια μεγάλη διάχυση χρειάζεται σχέδιο πολύ συγκεκριμένο το οποίο θα πρέπει να συνταχθεί με τη δέωσα επιμέλεια, να συζητηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το σχέδιο της κάθε χώρας πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις σχετικές διαστάσεις. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, είναι όμως εφικτό. Πρέπει κανείς να συνδυάσει τα κονδύλια από την παράταση με το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση ουσιαστικά παρατείνει τη χρονική ε, προθεσμία για να χρησιμοποιήσει μια χώρα τα εθνικά κονδύλια που της αναλογούν από τα ευρωπαϊκά και συνδυάζει τα εθνικά κονδύλια και ε, τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής. Βασιζόμαστε στα συνήθεια εργαλεία χρηματοδοτικά που μας δίνει η πολιτική συνοχής θα στηρίξουμε δηλαδή την απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους εργαζόμενους, θα στηρίξουμε τη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης, θα, δώσουμε, θα στηρίξουμε την παροχή ε, κινήτρων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα στηρίξουμε την δημιουργία νέων επιχειρήσεων τύπου, από αποφύτους πανεπιστημίων, για παράδειγμα, ε, προκειμένου να, υπάρχει, να υπάρξει επιχειρηματικότητα. Θα έχουμε την πολιτική των ανοιχτών θυρών, προτεραιότητα για το EU Invest και άρα μπορεί κανείς να διαπραγματευτεί project τα οποία θα τύχουν πολύ πιο εύκολα χρηματοδότησης από την τράπεζα, π.χ. αναδιάρθρωση του συγκεκριμένου κλάδου, της συγκεκριμένη βιομηχανίας που είναι παρούσα στην περιοχή ή χρηματοδότηση και με τραπεζικό δανεισμό ε, τεχνολογικών οικονομικών δραστηριοτήτων ή ε, δραστηριοτήτων που συνδέουν αυτή την περιφέρεια με άλλες ε, περιφέρειες έτσι ώστε να υπάρξει ομαλή ανάπτυξη. Δηλαδή τις λεπτομέρειες θα τις ρυθίσουμε στη συνέχεια, αλλά μιλούμε κατά βάση ε, δημόσιες υποδομές. Για τέτοιου είδους δημόσιες ε, υποδομές έχουμε το εργαλείο ε, για το χρηματοδοτικό της χρηματοδότησης τραπεζικής που στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη περιφερειακή διάσταση, τους ώστε να έχει νόημα αυτό το σχέδιο και μετά πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες. Προς τα πού θέλουμε να πάμε, ποια θα είναι τα σημεία αγκίστρωσης, αν θέλετε, τα ε, σημαντικά κατόφλια που θα πρέπει να φτάσουμε για να περάσουμε στην ανάπτυξη των περιφερειών και ποια θα είναι η προσέγγιση από τη βάση της πυραμίδας προς τα πάνω, από χαμηλά προς τα ψηλά. Πρέπει οι περιφερειές με το κράτος, το εκάστοτε κράτος να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ε, δουλέψουν σοβαρά για την υποβολή σχεδίου. Δεν γίνεται μία νυχτή, δεν γίνεται ω εκθαύματο. Α ασχοληθούμε, ας κόσουμε τα μανίκια, να ασχοληθούμε με το μέγιστο αυτό θέμα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να κομίσω. Ευχαριστώ ο Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ και θα συμπληρώσω λέγοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να αναλάβει πλήρως το ρόλο του συνομοθέτη που του αναλογεί. Και η δική μας Επιτροπή για τις Περιφέρειες έχει φτάσει στο μέγιστο σημείο κινητοποίησης για την νομοθετική διαδικασία. Ολοκληρώνεται ο πρώτο γύρο τραπέζης. Έχουμε ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο κατά τον οποίο δώσαμε το λόγο στους βουλευτές. Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Νίκο Ρώση, πρόεδρο της Περιφερειάς της Τοσκάνης και αντιπρόεδρο της CRPM, της Επιτροπής της Ένωσης των ε, Περιφερειακών ε, Εδαφών και Επικρατιών και ε, της Ευρώπης. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον συνάδελφο Ενρίκο ε, Ρώση, πρόεδρο της περιφέρειας της Τοσκάνης, περιφερειάρχη δηλαδή, πριν ε, ξεκινήσει επόμενος ε, γύρος με τους ομιλητές. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε. Είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί η φωνή των περιφερειών σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή. Θα ήθελα να πω εξ αρχής ότι συμφωνώ με τις σκέψεις της Επιτρόπου Φερέιρα όταν λέει ότι οι πολιτικές συνοχής θα πρέπει να ενταχθούν στις περιφερειακές συγχρηματοδοτήσεις καθώς και τις κρατικές χρηματοδοτήσεις για την οικολογική σύγκληση, για το πράσινο σύμφωνο και για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Πρόκειται για μια ε, πολιτική αλληλοσυμπλήρωσης. Αλλά θα ήθελα να εκφράσω και ορισμένες ανησυχίες. Μιλάμε για επιπρόσθετα 7,5 δις. Είναι πραγματικά επιπρόσθετα ή θα δούμε περαιτέρω περικοπές στην πολιτική συνοχή σε σχέση ε, με αυτά που προϋπόθηκαν. Ο πρόεδρος μας είπε κάτι το πολύ σωστό. Ποιος υποστηρίζει τις πολιτικές συνοχής. Αυτά τα χρήματα προς τις περιφέρειες θα πρέπει να εντάσσονται στο Green Deal, δηλαδή υπέρ της έρευνας ε, και της γεωργίας καθώς και της κατάρτισης. Θα πρέπει να υπάρχει αυτή η άμεση αιρεσιμότητα. Εάν λοιπόν αρθούν ή αφαιρεθούν χρήματα από την πολιτική συνοχής, δεν θα είναι επαρκής η χρηματοδότηση στο τέλος. Αυτό είναι κεφαλαιόδους σημασίας γιατί γίνεται λόγος για νέο χρήμα, αλλά από πού θα λάβουμε αυτά τα χρήματα. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν ε, ε, δεσμεύσεις που θα πρέπει να ξανασυζητηθούν σε σχέση με την οικολογική μετάβαση, δηλαδή να υπάρχει και ένα πλαίσιο φορολόγησης. Η ομάδα Μόντι ακριβώς ασχολήθηκε με αυτό, έτσι ώστε να υπάρχουν ανεξάρτητες ε, χρηματοδοτήσεις. Τέλος, πιστεύω ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Αυτό είναι απαράβατο, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε τους κινδύνους υποτίμησης των επιπτώσεων αυτής της ε, μετάβασης στην απασχόληση, στο χώρο εργασίας. Δεν είναι ιδιαίτερα απλό. Ή η μετάβαση θα είναι ρυθμιζόμενη ή όπως έγινε και με την παγκοσμιοποίηση, δυστυχώς ε, θα πληρώσουν το τίμημα, θα πληρώσει το τίμημα η εργατική τάξη. Εδώ μιλώ για τους ανθρακορίχους, αλλά και για τους εργαζόμενους στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Πώς θα υπάρχει δίκαιη μετάβαση. Ε, θα υπάρξει επαρκής ε, χρηματοδότηση στα πλαίσια της κατάρτισης ή χρειάζονται ε, νέα μέσα. Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να απαντήσετε τώρα κύριε Επίτροπε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις σας. Το πρώτο που είπατε σχετίζεται με το γεγονός ότι πράγματι χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους στον προϋπολογισμό. Ναι, είναι η απάντηση σε αυτό. Και ναι, χρειαζόμαστε και νέους πόρους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει μέρος του φο... των εισοδημάτων, των εσόδων από το φόρο για τον άνθρακα μπορεί να μπει στους ίδιους πόρους και είναι ένα ζήτημα που έχει μπει στην ημερησία διάταξη ή θα μπορούσε να μπει, δεν ξέρω αν ήσασταν ε, προηγουμένως όταν το είπα. Είναι αδύνατο. Με αυτό το επίπεδο ολοκλήρωσης της Ευρώπης και ένωσης, με αυτό το επίπεδο εσωτερικών αποκλήσεων με βάση τον ανταγωνισμό, να παραμένουμε με ένα προπολογισμό της τάξης του 1% και να συζητούμε ατέρμονα αν πρόκειται για 1,7, 1,07, 1,3, 1,0 κάτι. Δεν είναι δυνατόν. Είναι δυσανάλογα μικρό με αυτό το επίπεδο ολοκλήρωσης στο οποίο έχουμε φτάσει ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν μια συζήτηση η οποία αφορά όλους τους Ευρωπαίους, θα πρέπει όλοι να συμμετάσχουν και μάλιστα να εθετήσουν λόγο ειλικρινή. Θυμάμαι πολύ καλά την πρόταση του Μάριο Μόντι και είχαμε μιλήσει για κείμενο για το χρηματοπιστωτικό τομέα, για φόρο σχετικό για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Μιλήσαμε για φορολογία για τη χρήση πλαστικών. Υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικέ για να υπάρξουν περισσότεροι ήδη οι πόροι. Όμως και μεγαλύτερος να είναι ο προπολογισμό πρέπει να κινητοποιηθούν ιδιωτικοί πόροι για να προχωρήσει το πράγμα. Από εκεί και πέρα η παρουσία της Ευρώπης σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλανήτη, το πώς θα ρυθμίζουμε τα θέματα με τρόπο ώστε να μην σημειώνεται απώλεια θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη ε, και πώς θα γίνεται να ε, το ρηπογόνο κομμάτι της, βιομηχα... της οικονομίας να το απολέσουμε. Εγώ για πάρα πολλά χρόνια είμαι Πέρι της εξής άποψης, να έχουμε benchmark σημεία αναφοράς ανακλάδο και αυτά τα σημεία αναφοράς να τύχουν συμφωνία σε διεθνές επίπεδο και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ λεπτομερές αυτό το εγχείρημα. Ακόμα και αν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν αναλάβουν τη δέσμευση ότι σε όποια τεχνολογία και αν ε, καταλήξουν και εφαρμόζουν σε ό,τι έχει να κάνει με το αντίκτυπο για το κλίμα εντός, στο εσωτερικό τους, άρα στην Ευρώπη, θα την επιβάλλουν αυτή ε, θα την επιβάλλουμε αυτή και στους υπεργολάβους και στους αναδόχους με τους οποίους συνεργάζονται σε τρίτες χώρες. Και αν δεν την επιβάλλουν και οι άλλες επιχειρήσεις να τη χρησιμοποιούν στις χώρες και τις περιφερειές τους, το μόνο τελικά που θα κάνουμε είναι να εξάγουμε θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργούνται αλλού δηλαδή εκτός Ευρώπης, αλλά να εξάγουμε και μόλις η ρήπανση η οποία θα σημειώνεται αλλού. Ε, Πρέπει ε, να έχουμε αυτές τις καλές προθέσεις, να μην καταλήξουμε τελικά να εξάγουμε θέσεις απασχόλησης και να εξάγουμε ρήπαση. Απλά να, τη μεταθέτουμε, να μην γίνεται στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, αλλά να γίνεται αλλού. Αυτά πρέπει να τα προσπαθήσουμε και για το καλό του πλανήτη, όχι μόνο για το καλό των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Έχουμε 15 ε, συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ζητήσω από όλους σας να είστε συνοπτικοί, να είστε συγκεκριμένοι στα ερωτήματα που θα θέσετε. Ο Πέντρο Μάρκες από τους Σοσιαλιστές, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω πορτογαλικά, που είναι και η μητρική γλώσσα της Επιτρόπου και η δική μου. Αγαπητή Επίτροπε, αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για εμένα που θα συνεργαστούμε κατά την επόμενη πενταετία και πιστεύω ότι η κοινή μας εργασία θα στεφθεί από επιτυχία. Τουλάχιστον θα το προσπαθήσουμε. Η Κωνσταντς Κρέλ έθιξε ένα από τα ζητήματα που μας απασχολούν όλο ένα και περισσότερο, δηλαδή η μετάβαση πόρων σε χώρες ή περιφέρειες που θα έχουν μεγάλα προβλήματα στήριξης από το 2021 και θα θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με τον αποκλεισμό από πλευρά Συμβουλίου κατά παράδεκτο τρόπο. Οι συζητήσεις δεν μπορούν να συνεχιστούν ως προς το ΠΔΠ. Σε σχέση με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα ήθελα να πω ότι στο Πράσινο Σύμφωνο η Επιτροπή προέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις με νέο χρήμα στα πλαίσια του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Και όπως είπε και ο Περιφερειάρχης ε, από την Ιταλία, χρειαζόμαστε να υπάρξει απτή εφαρμογή, γιατί μιλάμε για επιπρόσθετα 7,5 δις, επιπροσθέτως δηλαδή από την πρόταση της Επιτροπής. Αν δεν ακούσουμε από το Συμβούλιο να λέει ότι δέχεται αυτή τη βάση διαπραγμάτευσης, δεν έχει νόημα να μιλάμε για νέο χρήμα. Θα θέλαμε αυτά τα νέα χρήματα να προέρχονται πέραν από την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μιλάμε για ίδιους πόρους για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και για νέο χρήμα επιπροσθέτως αυτών των πόρων. Αν δεν έχουμε αυτή την εγγύηση, τότε θα έχουμε μία ε, επικοινωνιακή πολιτική πολύ καλή, αλλά ως προς το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν μπορούμε να μιλάμε για νέο χρήμα, αλλά για συνεχείς απογοητεύσεις. Ένα δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να θίξω σε σχέση με το ρυθμιστικό πλαίσιο που θίξατε και εσείς οι ίδια. Υπάρχει ένα άνοιγμα συζήτησης και υπάρχουν στοιχεία που μας καλύπτουν, αλλά άλλα που μας ανησυχούν. Θεωρώ ότι φτάνουμε σε ένα γραφειοκρατισμό των περιφερειακών σχεδίων και μέσα στα πλαίσια αυτής της συνολικής εκτίμησης είναι πολύ δύσκολο να καταρτήσουμε περιφερειακά και εδαφικά προγράμματα τη στιγμή που πολλές περιφέρειες ε, μπορούν να καταρτήσουν αυτές, αυτή την οριοθέτηση χωρίς την επέμβαση της Κομισιόν. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μία ε, κοινή διαχείριση έτσι ώστε να αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Δεν έχει νόημα να έχουμε αυτή την ε, συγκεντρωτική προσέγγιση της Κομισιόν ως προς τη διαχείριση. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω το, το θέμα της διάρθρωσης του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Μπορούμε να ορίσουμε αυτές τις περιφέρειες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολύ φτωχές περιφέρειες οι οποίες δεν μπορούν να τύχουν χρηματοπιστωτικής υποστήριξης από τις μεγάλες τράπεζες. Θα πρέπει να ξέρουμε κατά πόσο υπάρχουν εγγυήσει έτσι ώστε να φτάσουν οι ιδιωτικές επενδύσεις στις πιο φτωχές περιφέρειες της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παπαδημούλης, παρακαλώ, αντιπρόεδρος. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καλωσορίζω την παλαιά συνάδελφο και φίλη Ελίζα Περέιρα στην Επιτροπή μας. Θυμάμαι μια φράση από την ακρόασή σας, αγαπητή κυρία Περέιρα, όταν ήρθατε πριν την έγκριση της Κομισιόν στην Επιτροπή μας. Επιβεβαιώνω ότι θα παλέψω στο Κολέγιο των Επιτρόπων για τον υψηλότερο δυνατό προϋπολογισμό. Εδώ είμαστε τώρα διότι η πρόταση της Κομισιόν είναι αδύνατο να χρηματοδοτήσει τους στόχους που η ίδια η Κομισιόν έθεσε. Απέχει πολύ από αυτά που ζητά με μια ευρύτατη πλειοψηφία το Ευρωκοινοβούλιο και ακόμη χειρότερα το Συμβούλιο ζητά δραστική περικοπή και αυτών που προτείνει η Κομισιόν που κατά τη γνώμη μας είναι ισχνά ανεπαρκή για να υπηρετήσουν την κοινωνική και την περιφερειακή συνοχή. Και επειδή ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις, αλλά οι αριθμοί στο τέλος μετρούν, βλέπω ότι η πρόταση της Κομισιόν για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο έχει μείωση μείον 11% για την περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή ειδικά για το Ταμείο της Συνοχής μείον 45%. Για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μείον 7%. Και σας ερωτώ πώς θα υλοποιηθούν οι στόχοι που εσείς θέσετε με αυτά τα χρήματα. Τι θα κάνουμε για να αγωνιστείτε όπως μας υποσχεθήκατε μαζί μας για να ανέβουν αυτά τα κωδία. διότι τα χρόνια αυτά οι ανισότητες κοινωνικές και περιφερειακές αυξήθηκαν. Και δύο πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Όταν παρουσιάσατε το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, μας είπατε ότι τα 7,5 δις είναι φρέσκο χρήμα. Επειδή όμως οι μειώσει που προτείνει η Κομισιόν στις πολιτικές συνοχής είναι πάνω από 30 δις, μήπως δεν είναι φρέσκο χρήμα, αλλά απλώ εκεί πηγαίνει το 25% από τις περικοπές των πολιτικών συνοχής. Και η δεύτερη ερώτηση εκτός από τα κριτήρια που έχετε θέσει για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης. Θα βλέπατε να προσθεθούν και κάποια άλλα ζωτική σημασία κοινωνικά κριτήρια όπως είναι ο δείκτης της ανεργίας στη χώρα και στην περιφέρεια. Για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία είναι πάρα πολύ ψηλή η ανεργία. Ή η ηλικία αυτών που απειλούνται από την ανεργία. Για να είναι πιο δίκαιη κοινωνικά η μετάβαση. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Η Ιζαμπέλα Μπεντζεά, αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ, θα μιλήσω ισπανικά. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Καλώς ορίσατε. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που ζήτησαν το λόγο γι' αυτό και θα είμαι σύντομη. Θέλω πρώτα να εκφράσω μια σκέψη και μετά θα διατυπώσω ερώτηση. Είπατε ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή τη συζήτηση της παλιάς πολιτικής ε, πολιτική συνοχή, νέε πολιτικέ και ούτω καθεξής. Όμως η πολιτική συνοχή και η πολιτική περιφερειακή ανάπτυξη φαντάζει συχνά κάτι το μακρινό σε σχέση με τον Ευρωπαίο πολίτη. Δυσκολευόμαστε να την καταστήσουμε πιο ορατή και να κάνουμε τη σωστή επικοινωνία προ τον Ευρωπαίο πολίτη. Ε, υπάρχει αντίληψη ότι δαπανώνται πολλά εκατομμύρια ευρώ τα οποία βγαίνουν από του φόρου που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι και συνεχώ μιλούμε για τη διευκόλυνση, τα, με μεγέθυνση και τη διεύθυνση αυτού του προϋπολογισμού. Υπάρχει πραγματικός αντίκτυπος, μπορούμε να μιλήσουμε για συγκεκριμένα πράγματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα. Ποια μέτρα έχετε για να ε, στηρίξετε την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ήπεθρο. Ποια μέτρα θα καταστήσουν δυνατό π.χ να ε, πληρώνεται μια μικρομεσαία επιχείρηση σε διάστημα μικρότερο των 90 ημερών από το κράτος. Γιατί στην Ισπανία σήμερα τουλάχιστον τρει μήνες, τουλάχιστον 90 μέρες πρέπει να περάσουν για να πληρωθεί κάποιος προμηθευτής. Πώς μπορούν να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις στην Ισπανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ε, γίνει αυτή η πολιτική συνοχή, να υπάρχει ορατότητα, να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα. Και Συμφωνώ με την ε, όλη νοοτροπία του Ταμείου για τη, δίκαιη, για τη μετάβαση. Δεν θα επεκταθώ γιατί ήδη το έχουμε αναλύσει σε βάθος σήμερα το πρωί. Ο Πρόεδρος Πασκάλ Ριμπον, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ. Και εγώ θα ήθελα να σας ε, ε, ευχηθώ ό,τι καλύτερο και κυρίως υγεία για το 2020 και θα ήθελα να πω ότι στη τελική ανάλυση ο πολίτη θα τα νιώσει όλα αυτά στον τραπεζικό του λογαριασμό. Αυτό είναι το θέμα στην τελική ανάλυση. Ό,τι όμορφο και να λέμε, ό,τι ε, κείμενα νομικά και να γράφουμε, όσο ακριβή και αν είναι, αν σε τελική ανάλυση είναι πίσω ε, στην τράπεζά τους ε, κάθε μήνα, όλα αυτά θα είναι άσχετα. Το Συμβούλιο κάνει ωραίες ομιλίες κάθε φορά και κάθε φορά προεξαγγείλει ε, το πράσινο, την πράσινη συμφωνία. Αλλά όλα αυτά χρειάζονται χρήματα. Εδώ χρειάζονται αναδιαστρώσεις, αλλά θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις, να επενδυθούν χρήματα. Στην παρούσα φάση είμαι πεπισμένο ότι αν το κλίμα ήταν τράπεζα θα το είχαμε σώσει εδώ για καιρό. Και θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πιο συγκεκριμένοι πιο λεπτομερείς και ξεκινάμε από την πολιτική συνοχή, γιατί η πολιτική συνοχή είναι κομμάτι της νέας πράσινης συμφωνίας. Αν το Συμβούλιο όλα αυτά μέχρι τέλους 2020 ε, τα αναβάλει και τα ξαναβάλει, θα την πληρώσει όχι μόνο το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θεωρώ ότι την πλευρά μας, αλλά κυρίως θα πονέσουν οι χιλιάδες δικαιούχοι της πολιτικής αυτής. Αν θέλουμε να αποτρέψουμε την ε, περαιτέρω επιδείνωση του κύρου της Ευρώπης, θα πρέπει να μην ακολουθήσουμε αυτό που προτείνει και αυτό που έχει σκοπό να κάνει το Συμβούλιο. Αυτό το λέω ευθύ εξ αρχής για τα ζητήματα τα οποία συζητήσαμε σήμερα. Να μην επανέλθω γιατί πολλά ακούσαμε, αλλά τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις επιτρέψτε μου. Στην παρούσα φάση η πολιτική συνοχής έχει ζήτημα γιατί το ποσοστό απορρόφησης ε, των πόρων είναι αρκετά κακό. Αν θέλουμε να συγκεντρώσουμε περαιτέρω επιχειρήματα για να πείσουμε το Συμβούλιο, θα πρέπει να βελτιωθεί το ποσοστό απορρόφησης. Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε προς την κατεύθυνση αυτή. Και αυτό συνδέεται και με το μελλοντικό GTF για το Ταμείο Δίκαιης ε, Μετάβασης. Ε. Πώς μπορούμε λοιπόν να διδαχτούμε για να διαμορφώσουμε καλύτερα και τα θέματα αυτά. Ένα τεχνικό τώρα ζήτημα για την πρόταση για το Ταμείο Δίκαιης ε, Μετάβασης. Εδώ πέρα η Επιτροπή προτείνει να εξαιρεθούν τα στοιχεία τα οποία δεν εμπίπτουν την Πράσινη Συμφωνία και τα αρκετά καύσιμα, συμφωνώ, αλλά αποκλείονται και υποδομές για αέριο. Εγώ είμαι πεπισμένο ότι αν θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μετάβαση, το υδρογόνο αποτελεί βασικό και κρίσιμο στοιχείο για να πετύχουμε αυτή τη μετάβαση και χρειαζόμαστε υποδομές για τη μεταφορία του υδρογόνου. Έχουμε λοιπόν υποδομές για το αέριο σε πολλές χώρες, πολύ απλά θα χρειαστεί μία μετατροπή. Γι' αυτό χρειάζονται πόροι. Δεν έχει λοιπόν νόημα, θεωρώ, να εξαιρεθούν αυτές οι υποδομές από την επιδότηση. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω για ποιο λόγο εξαιρούνται και αποκλείονται τέτοιες επενδύσεις. Ευχαριστώ, Πασκάλ. Και βλέπω ότι αναφέρεται και υπάρχει καλή εκπροσώπηση. Να δώσω το λόγο στους, ε, στους πράσινους. Στον κύριο Ροπέ. Euh, Αν μου επιτρέπετε, ε, ευχαριστώ Πρόεδρε και κυρία Επιτροπέ. Μία πρώτη ε, ερώτηση. Είμαι από την Κορσική και είμαι από τους ε, βουλευτές που απασχολούνται πάρα πολύ για το θέμα των νησιών. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποκλείσει τη δυνατότητα συγκεκριμένη ε, ε, επικέντρωση και σε νησιωτικέ περιοχέ. Ωστόσο, αυτό αποτελεί μια ανάγκη, ιδιαίτερα ε, δεδομένη τη πολιτική προτεραιότητα για την οικολογική επικέντρωση στι περιοχέ, που είναι οι περιοχέ που έχουν τη μεγαλύτερη χρήση άνθρακα. Και η Νέα Επιτροπή και εσεί ιδιαίτερω θα ήταν σε να ξανακοιτάξει το επιχείρημα αυτό προκειμένου η Ευρώπη να δώσει με πιο μεγάλη σημασία στις νησιωτικές περιοχές. Δεύτερη ερώτηση, αν με επιτρέπετε, το ψήφισμα που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης αναφέρει συγκεκριμένα τα θέματα των περιφερειών στη σύνθεσή της και μου προκαλεί ε, εντύπωση αυτό, γιατί αυτό δεν συνήθιστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα αποδεχόταν την προσωπία των ε, περιοχών αυτών στην διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Φρανσουά, λέει ο Πρόεδρος και το λόγο τώρα έχει η συνάδελφος κυρία Μόσκα, αν είναι ακόμα στην αίθουσα. Δεν τη βλέπω. Μόστανόφσκα ονομάζομαι, λέει η κυρία Μόστανόφσκα. Να διορθώσω λοιπόν την προφορά του Ευχαριστώ, Επιτρόπε, και σας εύχομαι κάθε επιτυχία για το νέο έτος. Από πλευράς προπολογισμού θα είναι δύσκολο το έτος. Είπατε σε κάποια φάση ότι πρόκειται να προασπιστείτε την πολιτική συνοχή και αυτή την αρχή εταιρική σχέση. Ελπίζουμε, ελπίζουμε αυτή η υπόσχευση να τηρηθεί. σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή και το Ταμείο Πολιτική Μετάβαση. Ελπίζουμε να μην μείνουν καμία περιοχή. Και επίση, μα ε, υποσχεθήκατε να ενισχυθεί η πολιτική συνοχή στην περίοδο μετά το 2020. Έχουμε τεράστιε προκλήσει σε ό,τι αφορά το κλίμα. Επ' αυτού όλα συμφωνούμε. Υπάρχουν και πολλά αμφιλεγόμενα ζητήματα όμω. Το ύψο των πόρων, το πώς θα γίνουν οι εκχωρήσεις, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες για τη χρηματοδότηση και θα ήθελα να επανέλθω στο ερώτημα που έθεσε ο προηγούμενος μελητής. Η περιβαλλοντική ουδετερότητα. Το Συμβούλιο, όπως και η κυρία Επιτροπός, υπογράμμισαν το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη έχουν σημείο αφετηρίας διαφορετικό και θα πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν για το ενεργειακό τους μείγμα γιατί λοιπόν αποφασίσατε να περιορίσετε το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και γιατί εξαιρείτε τις ε, υποδομές αερίου από τις επιδοτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ξέρω, ξέρω πόσο δυσάρεστο είναι όταν κανείς δεν προφέρει καλά το σωστά το όνομά του, γιατί συμβαίνει και σε εμένα, ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος μιλητής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα όσα είπατε γιατί εκφράσατε πολύ σωστά το όλο πλαίσιο. Νομίζω ότι υπάρχουν χώρες που θέλουν να κάνουν περισσότερα με λιγότερα, με λιγότερα χρήματα. Δεν μπορούμε να προβάλλουμε μία αγροτική πολιτική, πολιτική συνοχής επιβαρύνοντας τους αγρότες ή τις μειονεκτούσες περιφέρειες. Αυτό το ζει η χώρα μου, η Ρουμανία, σε σχέση με το τομέα της ε, μετανάστευσης. Και γι' αυτό θα πρέπει να παρέμβει η πολιτική συνοχή, η οποία πρέπει να είναι και υλοποιήσιμη, χωρίς πραγματική απλούστευση της διαδικασίας και για τις ΜΜΕ και τις τοπικές αρχές, έτσι ώστε να προβάλλουν θέσεις εργασίας που να είναι καλοπληρωμένες, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Διαφορετικά, οι άνθρωποι δεν θα παραμείνουν σε αυτές τις απομακρυσμένες περιφέρειες θα απεριμωθούν αυτές οι απομακρυσμένες περιφέρειες εάν δεν βρίσκουν οι νέοι ικανοποιητική εργασία. Ένα δεύτερο πρόβλημα που έχουμε εμείς είναι ότι δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό. Κυρία Επίτροπε, μίλησα με τον ε, αρμόδιο υπουργό και του είπα ποιο είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα και μου είπε το εξή. Οι επιχειρήσεις που έχουν απορροφήσει στα κοινοτικά κονδύλια δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Δεν βρίσκουν εργαζόμενους για την πραγματική απορρόφηση. Εμείς λοιπόν βλέπουμε ότι το εργατικό μας δυναμικό αποστραγγίζεται. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ως προς αυτό. Τώρα, ως προς τα ορυκτά καύσιμα. Είναι πολύ ωραίο να μιλάμε για εναλλακτικές πηγές ενέργειας και ούτω καθεξής. Εμείς έχουμε περιοχές που έχουν πολλά ανθρακοριχεία και δεν μπορούμε να τα καταργήσουμε δια Είναι πολύ δύσκολο να υποστηρίξουμε νέες τεχνολογίες. Δεν μπορούμε να προβάλλουμε νέες τεχνολογίες σε αυτές τις περιφέρειες. Γι' αυτό θα πρέπει να μου πείτε πώς μπορείτε να ε, συνδράμετε για να λυθεί το θέμα της έλλειψης εργατικού δυναμικού στις απομακρυσμένες περιφέρειες. Ευχαριστούμε πολύ. Η συνάδελφος Σουσάννα Περέσε ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας καλωσορίζω κυρία Επίτροπε. Νομίζω ότι το θέμα της δίκαιης μετάβασης είναι πολύ σημαντικό για την απομάκρυνση από τη χρήση του άνθρακα. Θεωρώ όμως ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις σε περιφέρειες οι οποίες καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες μείωσης εκπομπών του άνθρακα. Η Ισπανία κλείνει και τις ε, θερμοδυναμικές μονάδες αλλά και πολλά ορυχεία αλλά χάνονται πολλές θέσεις εργασίας και υπάρχει και απερίμωση περιφερειών. Ξέρετε ότι η Ισπανία βρέθηκε σε δινή θέση σε σχέση με τη χρήση του Ταμείου δίκαιης μετάβασης. Χάθηκαν πολλές θέσεις εργασίας σε αυτή την περιοχή. Αυτό που με εκπλήσει ως προς τον μηχανισμό είναι ότι η λήψη των ε, πόρων δεν συνδέεται άμεσα με τους στόχους ε, αποσόβησης κινδύνων κλιματικής αλλαγής. Έχει λοιπόν σημασία να πρημοδοτήσουμε τις περιφέρειες οι οποίες πραγματικά προβαίνουν στη σωστή στοχοθέτηση. Τέλος, μας απασχολεί το θέμα των καθυστερήσεων των διαπραγματεύσεων για το ΕΤΠΑ, διότι μέσα στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ΕΤΠΑ και έτσι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να προετοιμάσουν τα επιχειρησιακά σχέδια για τις ΜΜΕ και για όλες τις επιχειρήσεις. Θα θέλαμε να οριστεί τελικά το ΠΔΜ ΠΔΠ με συγχωρείτε, το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε πολύ η Ρόζα Νταμάτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο. Καλώς ορίσατε. Εγώ θα ε, σταθώ σε ερωτήσεις και μόνο. Οι, οι, οι τρεις πυλώνες του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης είναι το μέσον μόχλευσης το οποίο έχει υπερτιμηθεί. Έτσι βλέπουμε ότι θα πρέπει να ενδυναμώσουμε όλες αυτές τις συνιστώσεις έτσι ώστε αυτό το carbon tax να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί γιατί και ε, το WWF μιλάει για χρήματα υπέρ του κλίματος τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα πράσινων επενδύσεων, κάτι το οποίο σέρνουμε από την προηγούμενη θητεία μας. Στη συνέχεια, πώς χρηματοδοτείτε αυτό το ταμείο. Πολλοί μίλησαν για το αέριο. Θα ήθελα να σας πω ότι πρόκειται για συγκεκριμένο ορυκτό καύσιμο. Και γι' αυτό νομίζω ότι δεν είναι και ο απότερος στόχος του Ταμείου. Η Επιτροπή, η προηγούμενη Επιτροπή προσέδωσε 29 ε, δις για τους αγωγούς. Δεν χρειάζεται λοιπόν να χρησιμοποιηθεί νέο δημόσιο χρήμα των Ευρωπαίων φορολογούμενων για μία άλλη πηγή. Γιατί ως προς το υδρογόνο και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας μπορούν να γίνουν πολλά. Τέλος, εγώ προέρχομαι από το Τάραντο που έχει τη μεγαλύτερη μονάδα χαλιβουργίας. Μιλώ για την Ήλβα. Και θεωρώ ότι θα μπορούσατε να μιλήσετε για μετατροπή ή κλείσιμο μονάδων που ενέχουν την χρήση των ορυκτών καυσίμων ή άλλων εκπομπών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι ακριβώς κάνουμε. Μιλάμε για μία μονάδα η κλεισιμο μοναδων που ενεχουν την χρηση των ορεικτων καυσιμων η αλλων εκπομπων θα πρεπει λοιπον να δουμε τι ακριβως κανουμε μιλαμε για μια μοναδα η οποια είναι ρηπογόνα. Καταρχήν σκοτώνει τους εργαζόμενους, για να μην μιλήσω για τους πολίτες. Εδώ και 50 χρόνια σκοτώνει τους ίδιους τους εργαζόμενους. Εγώ μιλώ από το κίνημα πέντε αστέρων και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ασφιχτιούν και άλλοι οικονομικοί τομείς. Εσείς θα πρέπει να βοηθήσετε ε, την δράση έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταργήσουμε αυτές τις χαλιβουργικές μονάδες, να προβούμε σε ένα ουσιαστικό decommissioning. Γιατί δεν μπορείτε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο και αυτή την μεγάλη έδρα της χαλιβουργίας που έχει μεγάλες επιπτώσεις κυρίως στο τομέα της υγείας. Διαφορετικά στο Τάραντο θα συνεχίσουν να πεθαίνουν άνθρωποι, να λιμοκτονούν και να πεθαίνουν κυρίως για λόγους υγείας. Ευχαριστώ πολύ. Άλβαρο Άλμερο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ, κυρία Επίτροπε, δεν είναι συχνές οι ευκαιρίες που έχουμε για να διαπιστώσουμε σύμπτωση απόψεων στα πλαίσια αυτής της διαλεκτικής μας πορείας. Εσείς όμως έχετε την αμέριστη υποστήριξή μας. Υπάρχει αλληλεγγύη στο Διευθυντήριο των Επιτρόπων, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό αλλά γνωρίζω ποιες είναι οι πεπιθήσεις σας και οι δυνατότητές σας για να μπορέσετε να ε, δράσετε έμπρακτα. Υπάρχει μία συγκεκριμένη αδιάσυστη πεποίθηση σε επίπεδο ευρωβουλευτών ότι πρόκειται για νέο χρήμα. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν μπορούν να αντιληφθούν πώς η Ευρώπη θέλει περισσότερη συνοχή και δεν προβάλλει το σωστό χρηματοοικονομικό πλαίσιο. Δηλαδή μιλάμε για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, αλλά μετά γίνονται ε, λιγότερες χρηματοδοτήσεις, λιγότερη χρηματοδότηση σε περιφέρειες που τη χρειάζονται περισσότερο. Δεν ξέρω κατά πόσο διατίθεται ακόμα λιγότερο χρήμα από τον ε, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για αυτές τις ε, περιφέρειες. Δηλαδή, οι πιο πλούσιες περιφέρειες λαμβάνουν περισσότερα. Αυτό εγώ βλέπω. Γιατί λοιπόν να μην υπάρχει ουσιαστική σύνοχη. Θα ήθελα να μιλήσω λοιπόν για την σωστή κατανομή στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ως προς την ε, άμεση ανάγκη επανόρθωσης. Μιλάμε για την ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο που θα πρέπει να κατέχει η ηγετική θέση στον κόσμο. Εμείς δεχόμαστε αυτό το σκεπτικό. Όμως δεν είναι δυνατόν να το κάνουμε αυτό, αλλά παράλληλα να μην σκεφτούμε τις περιφέρειες οι οποίες είναι οι πλέον αδύναμες, οι πλέον αποδυναμωμένες. Δεν μπορούμε με αυτή τη βαθμία προσέγγιση να εγκαταλείπουμε περιφέρειες που μας χρειάζονται. Και θα ήθελα στο μέλλον να λάβουμε υπόψη περιφέρειες που δεν παράγουν άνθρακα, αλλά που έχουν ε, και αντιμετωπίζουν πολλά δεινά, δηλαδή την απερίμωση. Δεν υπάρχει ζωή εκεί. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Εάν η Ευρώπη είναι διατεθειμένη για κάτι τέτοιο, για μία σωστή μετάβαση, τότε θα βοηθηθούν αυτές οι περιφέρειες οι οποίες δεν παράγουν άνθρακα, αλλά δυστυχώς βρίσκονται σε πολύ μειονεκτική θέση. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ήθελα όλοι σας να καταβάλετε μία προσπάθεια έτσι ώστε να υποβάλλετε σύντομες ερωτήσεις, διότι η Επίτροπος έχει να απαντήσει σε σωρία ερωτήσεων. Ο Κριστόφ Ζόρκελ έχει το λόγο. Ελπίζω να προέφερα καλά το όνομά σας. Αγαπητέ Πρόεδρε, κυρία Επιτροπέ, ποιος είναι ο στόχος της περιφερειακής πολιτικής. Μιλάμε για την ε, συνοχή. Και θέλετε να βοηθήσετε τις περιφέρειες που είναι οικονομικά ασθενέστερε. Αυτό διακηρύξατε. Χαιρόμαστε από πλευρά τη Πολωνία, γιατί μιλάτε για τις ε, περιοχές που είναι πίσω. Δεν ξέρω ποιες περιοχές όμως στην Πολωνία θα περάσουν αυτό το τεστ. Μιλάτε, για παράδειγμα, για την Ανατολική περιοχή της ε, Πολωνίας. Ενδεχομένως ε, η κυβέρνηση είναι σε ένα πρόγραμμα για την Ανατολική Περιφέρεια της ε, Πολωνίας. Μιλάμε για μια ομάδα των πέντε πιο ασθενών περιοχών στην Ευρώπη. Θα υπάρξει ειδική υποστήριξη για τις περιφέρειες αυτές. Γιατί νομίζω ότι πλουρούμε όλα τα κριτήρια που υπάρχουν. Και φυσικά το άλλο θέμα είναι πώς ορίζεται η δίκαιη μετάβαση, τι αποτελεί δηλαδή δίκαιη μετάβαση. Σας ευχαριστώ πολύ και το λόγο έχει η Σαμπέλα Κλοκ. Παρακαλώ σύντομη να είστε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Αγαπητέ Πρόεδρε. Όντως, ακούσαμε πολλές σημαντικές ερωτήσεις. Θα ήθελα να επαναλάβω όμως κάποιες πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Ποια θα είναι η πηγή των χρημάτων αυτό, αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια, από πού θα βγουν. Αναλυτικά θα θέλαμε να ξέρουμε. Υπάρχει αυτή η φοβερή καινούργια ιδέα, η πράσινη συμφωνία, πάρα πολύ φιλόδοξη, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι αναφορικά με το κλίμα. Πολύ ωραία. Αλλά βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια τι συμβαίνει και στις άλλες επίρους. Κάποια αριθμητικά στοιχεία επιτρέψτε μου να σας δώσω. από μια οργάνωση που παρακολουθεί την αγορά ενέργειας. Εντός 18 μηνών η Κίνα έχει αυξήσει την ενέργεια από άνθρακα κατά 40 γιγαβάτ. Ο κόσμος έχει μειώσει δε την αντίστοιχη ε, παραγωγή κατά 8,5 ε, κιλοβάτ. Έχουμε λοιπόν 37 γιγαβάτ ε, καθαρό πλεόνασμα. Αυτές είναι οι τάσεις. Δεν πρόκειται να αλλάξουν δε. Η Κίνα είναι σε φάση που ακόμα κατασκευάζει εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από άνθρακα σε ύψος 123 γιγαβάτ. Άρα, η δική μας προσπάθεια τι ακριβώς εξυπηρετεί σε ό,τι αφορά την ε, μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι λοιπόν. Και εγώ είμαι Πολωνή, ξέρω ποιο είναι το ενεργειακό μας μείγμα, όπως και όλος ο κόσμος. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, λοιπόν, αναρωτιέμαι, πρόκειται να παρέμβει. Θα προσπαθήσει να επηρεάσει το ενεργειακό μας μείγμα. Τη στιγμή που η συνθήκη προβλέπει κάποιες ελευθερίες. Έχουν αυξηθεί τα χρήματα από 4,8 δις σε 7,5 δις. Χαίρομαι. Αλλά να θυμάστε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της χώρας μας. Δεν μπορούμε να είμαστε ουδέτερη σε ό,τι αφορά το κλίμα μέχρι το 2050. Δεν μπορούμε να πετύχουμε την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Κατελίνη Ξέ ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και θα είμαι σύντομη. Επίτροπε. Την ε, προηγούμενη εβδομάδα Είσαστε από τους πρώτους όπου τονίσατε ότι ε, η ρεσιμότητα για το κράτος δικαίου θα ισχύει και για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Δεν ξέρουμε όμως πολλά σε ό,τι αφορά τον όρο αυτό του κράτος δικαίου. Διευκρινίστε παρακαλώ και σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις που αναλάβατε ως υποψήφια επίτροπος. Είπατε ότι δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι μεμονωμένοι δικαιούχοι των κάθε κράτους γιατί δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την κατάσταση σε ό,τι αφορά το κράτο στη χώρα τους ως Ούγγροι. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Πείτε μας λοιπόν, με ποιο μηχανισμό σκοπεύει να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλίσετε ακριβώ αυτό που υποσχεθήκατε, ότι δεν θα επηρεαστούν οι μεμονωμένοι δικαιούχοι, αλλά να υπάρχει περιορισμό τη απάτη. γενικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφο που είχε ζητήσει το λόγο από την Σοσιαλιστέ και Δημοκράτες. Ναι. Ευχαριστώ. Από το ECR. Κυρία Επίτροπε, έχουμε φιλόδοξα project, μεγαλειώδεις φιλοδοξίες πράγματι και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει αξιόπιστη ανάλυση πριν ξεκινήσει το κάθε εγχείρημα. Πόσο θα μας στοιχήσει αυτή η οικονομική μεταμόρφωση, ποιο θα είναι το εργασιακό κόστος, το κοινωνικό κόστος, πόσο θα υποφέρει ο κόσμος από αυτό το μεγαλειώδες εγχείρημα δεν θα έχουμε τεράστια αύξηση των ε, τιμών ενέργειας. Αυτό το είδαμε να συμβαίνει στη Γερμανία. Αναπάντητα παραμένουν αυτά τα ερωτήματα και οι ανάγκες στα κράτη-μέλη είναι τεράστιες, ειδικότερα στα κρατη που έχουν χαμηλό κατακεφαλήν εισόδημα σε σχέση με το ΑΕΠ, ε, όπως η Πολωνία, για χώρες που έχουν, ε, μεικτό, έχουν ενεργειακό μείγμα που έχει και τον άνθρακα μέρος του και λέγεται ότι οι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2030 και πρέπει 180 δις να επενδύεται ετησίως για να μπορέσει να γίνει αυτό εφικτό. Σε σύγκριση με αυτό το ποσό λοιπόν 7,4 δις στο Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση είναι ψίχουλα, είναι γελία τα χρήματα αυτά και τα κονδύλια αυτά αν μου επιτρέπεται ο όρος. Μιλούμε εδώ για την πίστοση, για τη χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τη χρηματοδότηση από τράπεζες και ούτω καθεξής. Το ταμείο αυτό δεν θα έχει κανένα αντίκτυπο για να γίνει δίκαιη μετάβαση. Γιατί η πόροι του είναι απειροελάχιστοι. Άρα, τι κρύβεται στο πίσω μέρος του μυαλού σας, ποια είναι ε, η αληθινή στόχευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναρωτιέμαι. Εμείς πηγαίνουμε ε, με 100 χιλιόμετρα, ε, οδεύουμε να προσκρούσουμε στο τοίχο της καταστροφής. Θα πλουτίσουμε τις τσέπες των πολυεθνικών που έχουν έδρα αλλού και θα πλουτίσουμε και τις τρίτες χώρες και τίποτα άλλο δεν θα γίνει και ορισμένοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν ήδη σε σημαντικά στατιστικά στοιχεία. Ήδη γίνονται τεράστιες θυσίε. Κάνουμε τεράστιες θυσίε. Η Πολωνία κάνει τεράστιες θυσίε, Αλλά σε σύγκριση με αυτό το οποίο συμβαίνει στην Κίνα, για παράδειγμα, αυτά που λέτε είναι έως και γελία. Ευχαριστώ η κυρία Κουταγιάρα από τους Σοσιαλιστές παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για τις παρατηρήσεις σας και για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ θυμάμαι την ακρόασή σας εδώ. Θυμάμαι ότι είπατε ότι κανείς δεν πρέπει να παραμείνει ε, στο περιθώριο, πρέπει να έχουμε συμπαράταξη και συμπόρευση και συμπερίληψη όλων των κοινωνικών ομάδων. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η δική μας Επιτροπή θα ασχοληθεί με μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για τη διάσταση του, των δύο φύλων σε σχέση με την πολιτική συνοχή. Είμαστε πολύ ευαίσθητοι στα θέματα της ισότητας των φύλων και του gender mainstreaming. Τα θέματα των φύλων δηλαδή να μπουν στο επίκεντρο οποιασδήποτε πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει τονιστεί επανειλημμένως η σημασία συγκεκριμένων εργαλείων, ύπαρξη συγκεκριμένων εργαλείων για να έχουμε μεγαλύτερη ισότητα και να ε, λαμβάνεται αυτό υπόψη σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Όλα αυτά είναι υποθέντα, λεχθέντα και γνωστά. Άρα, ποια βήματα έχετε πράξει, σε ρωτώ. Ε, τι έχετε κάνει διαφορετικό και πώς βλέπετε τις διαπραγματεύσεις για την περίοδο 2021-2027, για το πλαίσιο δηλαδή που θα ε, ε περικλείσει την πολιτική συνεχή... για το χρονικό διάστημα 2021-2027. Άρα, στη διαπραγμάτευση ρωτώ πώς έχετε λάβει υπόψη την ισότητα των φύλων, ε, την ενίσχυση των γυναικών και την φροντίδα των παιδιών. Έχετε τροποποιήσει ε, κάποιες πτυχές από το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για να μπει το θέμα των φίλων ε, σε όλες τις πολιτικές. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις έχουν ζητήσει το λόγο και κλείνει εδώ ο κατάλογος των ομιλητών που ζήτησαν το λόγο. Κόντε από το ID, Μέσρε Μαρτίν και Γκαρσία, Μουνιός. Αυτά. Δεν θα δώσουμε το λόγο σε άλλους. Παρακαλώ. Τρεις τελευταίοι ομιλητές. Καλημέρα σας κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που βρίσκετε βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων είναι πολύ σημαντική με βάση και τις επικείμενες διαπραγματεύσεις μετά το 2020. Πρόκειται για μια πολιτική που παρά το γεγονός ότι ήταν ευεργητική, έθεσε ένα αμφιβόλο το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου δυστυχώς θα υπάρξουν περικοπές κατά της περιφερειακής πολιτικής, χωρίς να υπόψη οι ανάγκες των περιφερειών, των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μία τέτοια προοπτική είναι ανησυχητική για μία χώρα σαν την Ιταλία, η οποία ε, βλέπει ότι μειώνονται δραστικά οι μεταβάσεις σε συγκεκριμένες ε, περιφέρειες καθώς και συγχρηματοδοτήσεις, ιδιαίτερα για το Interreg. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγήτρια για την σχετική έκθεση επίσης. Ε, δυστυχώς θα περικοπούν πολλά διαπεριφερειακά προγράμματα καθώς και διεθνικά. Εγώ εκπροσωπώ το Βένετο και τη ε, Βενέτσια Τζούλια, το βορειοδυτικό μέρος της Ιταλίας το Ιντερεγ βοήθησε στην εδαφική συνεργασία με τους γείτονες μέσω δεκάδων σχεδίων που επέτυχαν και που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στις όμορες περιοχές. Θα ήθελα λοιπόν σε σχέση με τις επερχόμενες περικοπές ε, να μπορέσει η Επιτροπή να υποστηρίξει το Interreg. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Μαστρέ Μαρτίνη, δύο σύντομες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, λέει η κυρία μαστρέ Μαρτίν. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για το ότι εκφράσατε και εσείς τις ανησυχίες μας. Αυτό που έχει σημασία είναι κατά πόσο μπορούμε να υπερβούμε τις δυσκολίες που υπάρχουν για την πρόσβαση στα ταμεία μετά την αναθεώρηση των κανονισμών. Οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η απλοποίηση, η απλούστευση, πώς μπορούμε να άρουμε τα προσκόμματα ως προς την πρόσβαση στα ταμεία. Όλα αυτά τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά και που όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι δεν μπορούμε πλέον να περιμένουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει αυτή η σύγκληση έτσι ώστε να μπορέσει κανείς να παρέμβει άμεσα. Πώς μπορούμε λοιπόν να άρουμε αυτές τις δυσκολίες, τι μπορούμε να κάνουμε με την απερίμωση των περιφερειών που μειονεκτούν. Μας ανησυχεί βεβαίως και το πράσινο σύμφωνο και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει για συγκεκριμένες χώρες θα πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία σε εγκάρσιο επίπεδο και αυτό αφορά όλες τις περιφέρειες. Ε, μην ξεχνάτε όμως ότι δεν ξεκινάνε από το ίδιο σημείο όλες οι περιφέρειες. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μεταχειριστούμε τα επιπρόσθετα αυτά κονδύλια για να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις και του Ταμείου Μετάβασης, γιατί στην περίπτωση της Ισπανίας υπάρχουν ε, ανθρακοφόρες περιοχές όπου έκλεισαν πολλά ορυχεία και θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραμείνουν ε, στις ευεργετούμενες περιφέρειες. Ε, ξέρω μία περίπτωση ε, ε, ενός ανθρακοριχείου το οποίο δεν έχει ε, κλείσει εδώ και πέντε χρόνια. Και βλέπουμε ότι μέσα σε πέντε χρόνια έχει προβάλλει μια διαφορετική απόδοση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει πραγματικά δίκαιη μετάβαση και κατά πόσο μπορείτε να το επιτύχετε αυτό. Ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις σας. Η συνάδελφος ε, Γκαρσία. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είχατε καταγράψει το όνομά μου πριν, αλλά φαίνεται ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ για τις επεξηγήσεις σας. Θα ήθελα να πω ότι το σχέδιο επενδύσεων ήταν πολύ καλό, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να υποστηρίξουμε τις περιφέρειες που προβαίνουν στην ενεργειακή μετάφαση, όπως η Αραγωνία, η δική μου περιφέρεια. Και βλέπω ότι υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις, επιπτώσεις οικονομικές και κοινωνικές, που θα μπορούσαν να έχουν ε, μεγάλες επιπτώσεις, ιδιαίτερα στο Ετερουέλ, γύρω στις 4.000 εργαζόμενοι εξαρτώνται από την εργασία στον τομέα του άνθρακα. Επίσης δεν μπορούμε να ξεχνάμε αυτούς οι οποίοι κατ έβαλαν κάθε προσπάθεια και έκαναν το δικό τους καθήκον. Θα πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν στην περιφέρειά τους, γιατί διαφορετικά γίνονται μετατάξεις που δεν ε, υπηρετούν κανέναν. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει επι, επι, απερίμονηση συγκεκριμένων περιφερειών. Υπάρχουν πολλά δημογραφικά προβλήματα και προκλήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και αυτό το κριτήριο στο Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης. Θα ήθελα να ξέρω, γίνεται κάτι τέτοιο, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε πολύ. Και φτάνουμε λοιπόν ε, στο τέλος ε, των ομιλητών μας. Δεν είναι εύκολη η δουλειά που έχετε να κάνετε, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα που ακούσαμε. Πραγματικά πολύ πολύ άριθμα. Έχετε λίγο πολύ 15 λεπτά στη διάθεσή σας για να απαντήσετε στις ερωτήσεις αυτές. Και να σας πω στο σημείο αυτό ότι έχετε ήδη δώσει απαντήσεις ε, στους συντονιστές και ενδεχομένω λοιπόν θα έχει νόημα για μας να ακούσουμε τα θέματα τα οποία δεν έχετε ήδη απαντήσει σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις που ακούσαμε και στο πρώτο τμήμα της συνεδρίασης. Έχετε το λόγο για 15 έως 20 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να συνοψίσω και να ομοδοποιήσω κάποιες από τις ερωτήσεις που ακούσαμε. Παρά το γεγονός ότι, όπως είπατε και εσεί Πρόεδρε, κάποιες ερωτήσεις έχουν ήδη ε, διευκρινιστεί και απαντηθεί για τα, το νέο χρήμα. Διάφοροι βουλευτές αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό. Ο, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να υποβάλει την πρόταση. Μετά οι συνομοθέτες είναι αυτοί που αποφασίζουν η πρόταση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν όπως έχω υποσχεθεί και στο παρελθόν, ήταν να εγγυηθούμε ότι θα προτείνουμε νέο χρήμα, 7,5 δις, το οποίο είναι ποσό ανώτερο των 4,8 δισεκατομμυρίων που είχε προτείνει το Κοινοβούλιο. Νέο χρήμα λοιπόν, πέρα από τις προτάσεις της προηγούμενης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχή το 2018. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε όλοι μας, αλλά πλέον οι συνομοθέτες είναι αυτοί που θα απαντήσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε την πρότασή της είναι κατά πάσα πιθανότητα η στιγμή να ασκήσουμε πιέσεις στα κράτη-μέλη, προκειμένου να προσεγγίσουν τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ προσωπικά αυτό που υποσχέθηκα είναι να αγωνιστώ για το πιο υψηλό δυνατό ποσό. Γι' αυτό αγωνίζομαι λοιπόν και νομίζω ότι είναι σαφές στην προτινόμενη ε, στον προτινόμενο κανονισμό ότι όλα αυτά είναι επιπλέον χρήματα. Αλλά όπως σας είπα, το μπαλάκι πλέον είναι στο γήπεδο των συνομοθετών. Εγώ θεωρώ ότι την υπόσχεσή μου την τήρησα. Δημήτρη, και εσύ το είπες, το είπαν και άλλοι βουλευτές. Σε σχέση με την ερώτηση του Πέντρο Μάρκες, τον οποίο θα ήθελα να χαιρετήσω. Σε σχέση με την μετάβαση μεταξύ ταμείων θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού και θα πρέπει να εγγυηθούμε να ε, υπάρξει μία ελάφρυνση του Συμβουλίου έτσι ώστε να δοθεί τελική μορφή στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, να μην δημιουργηθεί μεγαλύτερη αστάθεια με λίγα λόγια. Εμείς θα δεχτούμε αυτή τη στρατηγική συνεργασία επίσης. Προέκυψε το ζήτημα των ε, επενδύσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα στις διάφορες περιφέρειες. Έγινε λόγος για την ΕΤΕ και σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για τον τρίτο πυλώνα του της ΕΤΕ έτσι ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο των προγραμμάτων και γνωρίζουμε ότι το ζήτημα αυτό έχει συζητηθεί. Στόχος είναι κάθε επένδυση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης να αφήσει ανοιχτή πόρτα στις εγγυήσει των μέσων, έτσι ώστε αυτά τα προγράμματα να τύχουν προτεραιότητες, δηλαδή το EU Invest και το Ταμείο. Είναι ένα θέμα το οποίο σας απασχολεί και εσάς. Ε, ε, Δημήτρη, ευχαριστώ. Αλλά ήδη σας απάντησα. Σας απάντησα και προηγουμένως. Ως προς την ερώτησή σας θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ορατότητα από αυτή που ήδη έχουμε. Σας έδωσα πληθώρα παραδειγμάτων. Τώρα θα πρέπει να γίνει πίεση, να ασκηθεί πίεση προς τα κράτη-μέλη και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα ε, διαρθρωτικά ταμεία έτσι ώστε οι πολίτες να το αισθανθούν αυτό, να μην παραμείνει μια θεωρητική συζήτηση του κατά πόσο πρόκειται για 1,3, 1,7 θα πρέπει να εργαστούμε επιτόπου για να γίνει κατανοητό το όλο ζήτημα και από τους πολίτες και οι ευρωβουλευτές μπορούν να το κάνουν αυτό που γνωρίζουν τις περιφέρειες σε σχέση με την ερώτησή σας, κύριε Πασκάλα Ρημό. Το άκουσα και από άλλους συναδέλφους σας το ερώτημα αυτό, σε ό,τι αφορά το αέριο. Το Ταμείο Δίκης Μετάβασης έχει ως σκοπό να επιλύσει τα κοινωνικά προβλήματα, το θέμα της ε, ποικιλομορφίας και της, ε, της βιομηχανικής βάσης των ε, περιφερειών δεν αποσκοπεί στο αέριο. Το αέριο. Αν ε, χρησιμεύει στα περιφερειακά σχέδια, μπορεί να χρηματοδοτηθεί από, το, από τα περιφερειακά και τα εθνικά προγράμματα. Όχι από το Ταμείο Μετάβαση, γιατί δεν έχει νόημα, το είπε και ο συνάδελφο στην παρέμβασή του, ότι το αέριο ουσιαστικά δεν μπορεί να αποτελεί ε, κάτι το οποίο επιδοτείται έτσι, θα πρέπει να αποτελεί τμήμα ενός πακέτου το οποίο θα προωθηθεί από κοινό. Δεν είναι ο σκοπός αυτός του Ταμείου Δικής Μετάβασης. Ακούσαμε και ένα άλλο στοιχείο. Και συμφωνώ με τον συνάδελφο που ανέφερε, ο κ. Βούντο το ανέφερε, ότι υπάρχει ανάγκη απλοποίησης. Έχουμε καταβάλει εδώ ιδιαίτερες προσπάθειες για να απλοποιηθεί η όλη διαδικασία. Να δούμε κατά πόσον αρκεί αυτό. Αρκούν οι προσπάθειές μας. Θα το κρίνει το Κοινοβούλιο αυτό. Μα έλεγε ότι δεν υπάρχει ο κλιματικός στόχος. Υπάρχει όμως κλιματικός στόχος, υπάρχει αποφασιστικότητα επ' αυτού, γιατί είναι, συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο που καταρτίζουν τα κράτη-μέλη. Και αυτό το οποίο γίνεται είναι το εξής. Πρέπει μια περιφέρεια να είναι συμβατή με αυτό το σχέδιο. Το σχέδιο να καλύπτει μια περιφέρεια. Είναι απαραίτητο. Είναι καθοριστικό στοιχείο. Έτσι θα αλλάξουμε ε, τις εκπομπές ερήπων με την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου και στο Ζωζέ Νταμάτο έχω να απαντήσω για τις εκπομπές των αερίων και όντως για την ανάγκη να γίνει αυτή η μετάβαση είναι αναπόφευκτος, αναπόδραστος ο χαρακτήρας αυτή τη μετάβαση. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ETS, το σύστημα εμπορία εκπομπών ρήπων, ανταλλαγή και το, όλα τα ταμεία, τα κονδύλια για να ενισχύσουμε αυτή τη δουλειά έκανε ορισμένα σχόλια σε σχέση με αυτά που έχουν απαντηθεί. Τώρα, η περιφερειακή πολιτική δεν περιορίζεται στον μηχανισμό και στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Αφορά περιφέρειες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα. Και αυτό δεν σημαίνει ότι, δεν, ε, ότι καλύπτονται όλα, όλες οι πτυχές ε, της περιφερειακής πολιτικής. Και μετά είχαμε σχόλια από δύο συναδέλφους από την ε, Πολωνία. Έχω συνάντηση στην Πολωνία την επόμενη εβδομάδα. Δεν πρέπει να το βλέπετε ως μια επιβολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια ε, άνωθεν επιβολή. Είναι μια φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Όλοι προς τα εκεί πάνε. Προσπαθούμε να έχουμε ε, διάρκεια σε αυτές τις ε, δραστηριότητες. Και στην Ελλάδα υπόθηκε αυτό. Αυτές οι επιχειρήσεις χάνουν χρήματα κάθε μέρα. Άρα πρέπει να το πάρουμε απόφαση και να διαχειριστούμε τη μετάβαση αντί να υποκρινόμαστε ότι μπορούμε να σταματήσουμε τις αλλαγές και να έχουμε εσωστρέφεια. Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν και στην ε, και στην, ε, στα ναυπηγεία και στη χαλιβουργία. Ε, πρέπει απλά να διαχειριστούμε τη μετάβαση έτσι ώστε να μην απολέσουμε αυτονομία από πλευράς ενεργειακής και να μην δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα ε, για τον κόσμο και τους απασχολούμενους. Μπορεί να γίνει, το έχουμε κάνει και στο παρελθόν με άλλους κλάδους. Είμαι πολύ ευαίσθητη στα ζητήματα της ισότητας των φύλων. Θα πω στο τελευταίο λεπτό που έχω στη διάθεσή μου. Συζητούμε με τις υπηρεσίες ε, τι πρέπει να κάνουμε. Δεν θέλουμε να απλουστεύσουμε από τη μία ούτε να τα κάνουμε τα πράγματα υπερβολικά περίπλοκα από την άλλη. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή το μελωτούμε, πώς, ε, σε, με πιο σαφείς όρους θα α, εκπροσωπείται και θα παρουσιάζεται η ισότητα των φύλων στα κείμενά μας Νομίζω ότι έκανα μια φιλότιμη προσπάθεια να σας δώσω τις βασικές απαντήσεις, τα βασικά σας ερωτήματα. Είμαι διαθέσιμη και εγώ και οι συνάδελφοι και τα τμήματα και οι υπηρεσίες των οποίων προείσταμε να έχουμε ανοιχτό διάλογο μεταξύ, του, μεταξύ μας. Δεν λέω ότι είναι η καλύτερη δυνατή λύση, αλλά πρέπει τη μετάβαση να τη διαχειριστούμε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Δεν είναι κάτι το ιδανικό, είναι όμως κάτι απαραίτητο και γι' αυτό προσπαθούμε να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για όλους. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ο Πρόεδρος, κύριε Επίτροπε, εξ ονόματος του συνόλου των συναδέλφων, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω θερμά για τις πολύ συγκεκριμένες και ακριβείς απαντήσεις που μας δώσατε σε ερωτήσεις οι οποίες οφείλω να πω ότι όντως ήταν συγκεκριμένες και ακριβείς. Έτσι αντιλαμβανόμαστε τον απαιτητικό διάλογο υψηλού επίπεδου ε, που θα πρέπει να λαμβάνει η χώρα κάθε φορά που ε, έρχονται σε επαφή η δική μας Επιτροπή με τη δική, μας, με τη δική σας. Διαπιστώνω ότι σχεδόν τα περισσότερα ερωτήματα τέθηκαν για το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης. Αυτό δείχνει ότι η Επιτροπή μας έχει ε, κινητοποιηθεί σε αυτό το νομοθετικό και νομοπαρασκευαστικό έργο ε, για το οποίο θα συνεργαστούμε με εσάς. Και εσείς έχετε πολλά να κάνετε για αυτό το θέμα. Ο Άνθρακας είχε διαρθρώσει και δομήσει την ευρωπαϊκή οικονομία από τη βιομηχανική επανάσταση μέχρι και σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, κατά, τον, κατά τη γέννησή της ε, γεννήθηκε ως Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα άλλωστε. Επομένως, περιμένουμε με πολύ μεγάλη ικανοποίηση τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα επιδείξουμε τη δέουσα επιμέλεια για να βελτιώσουμε τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διαμορφώσουμε τη συζήτηση. Θα ήθελα να ζητήσω από τους διερμηνείς δύο λεπτά παραπάνω από το χρόνο τους για να μας βοηθήσουν έτσι ώστε να πω ότι προφανώς ε, όλα είναι τώρα, η μπάλα είναι στη πλευρά του γηπέδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό οι συντονιστές έλαβαν την απόφαση να αυξήσουν την πίεση που ασκείται ε, στο Συμβούλιο και είμαι σίγουρος κύριε Επίτροπε ότι και εσείς συμμερίζεστε την άποψή μου. Η πολιτική συνοχής δεν είναι πολιτική του παρελθόντος, δεν είναι πολιτική ε, πεπαλαιωμένη, παραδοσιακή. Ε, δεν τα, δεν βλέπω εγώ έτσι τα πράγματα. Η πολιτική συνοχή είναι μια ε, πολιτική του μέλλοντος, σήμερα που λαμβάνει η χώρα το Brexit, περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε την συνοχή. Είναι μια πολιτική η οποία έχει ήδη ε, διανύσει ε, αρκετή απόσταση σε ό,τι έχει να κάνει με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Στην περίοδο 2014-2020 κινητοποιήσαμε περισσότερα από 40 δις ευρώ για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της περιφέρειας, χωρίς να περιμένουμε το New Green Deal, τη νέα πράσινη συμφωνία της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπετε λοιπόν ότι είμαστε πρωτοπόροι. Θέλουμε να συνεργαστούμε για να εξυγχρονίσουμε ακόμα περισσότερο και να απλωστεύσουμε, όπως λέει και ο συνάδελφος Μπούντα, αυτή την πολιτική συνοχή έτσι ώστε η προστιθέμενη αξία Τη πολιτική αυτή, η οποία είναι ουσιώδης και πραγματική, να μπορεί επίση να γίνεται αντιληπτή από τον Ευρωπαίο πολίτη. Ίσως, κύριε Επίτροπε, έχει έρθει η ώρα να προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε σε σχέση με τη φιλανδική πρόταση τον προϋπολογισμό για άλλη μια φορά, συγκρίνοντας την και με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι σημαίνει αυτός συγκεκριμένα σε σχέση με... Ε, απώλεια έργων και δυσκολίες για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Να δούμε δηλαδή κάθε πρόταση πώς μεταφράζεται σε νούμερα και σε απώλειες για την πολιτική συνοχής. Να μην μιλούμε αυθαίρετα ή αν θέλετε